Καλό απόγευμα σε όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας λοιπόν. Ανακοινώσεις. Για την προηγούμενη μας συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο των συντονιστών ότι ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής ο κ. Διαμαντούρος ανακοίνωσε τη βδομάδα μας πέρασε την παρέτησή του που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την εκλογή του νέου διαμεσολαβητή. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το Σεπτέμβριο φέτος ώστε να μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος διαμεσολαβητής ε, την 1η Οκτωβρίου. Σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά και έκτακτες συνεδριάσεις μας που θα ορίσουμε όσο γίνεται συντομότερα και ασχοληθήκαμε με το θέμα του προγράμματος των διερευνητικών ε, αποστολών που είχαμε ορίσει από μερικούς μήνες πριν για την συνάντηση ας πούμε τη Μαδρίτη 22-23 Μαρτίου και το πρόγραμμα οριστικά υιοθετήθηκε επίσης στην Ελλάδα 28-31 Μαΐου το πρόγραμμα όμως που θα πρέπει να συμπληρωθεί με όσα θα μας πούν οι συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν τις υποδείξεις τους και περιμένουμε για να δούμε το πρόγραμμα της οργάνωσης της αποστολής στην Πολωνία που εκ νέου προσπαθούμε να οργανώσουμε να δούμε όμως πρώτα ποια θα είναι η σύνθεση της αποστολής της αντιπροσωπείας και ακόμα για την οργάνωση της δημόσιας ακρόασης 24 Σεπτεμβρίου την αποφασίσαμε στην Επιτροπή ΑΦΚΟ ακριβώς ε, μετά από την αναφορά για τα αποτελέσματα της ε, κρίσης της ε, οικονομικής ευρωπαϊκής πολίτες. Ήδη υπάρχει ένα πρώτο σχέδιο από τη Γραμματεία και τη δική μας και της ΑΦΚΟ και περιμένουμε να μας βοηθήσουν με υποδείξεις τα μέλη της Επιτροπής. Το είχαμε πει στην προηγούμενη συνάντηση ότι κάποιες αναφορές θα δείτε στο συνημένο έγγραφο ορισμένες ε, θεωρήθηκαν ε, μη παραδεκτές ε, λόγω αρχών και επιχειρημάτων συναδέλφων μας η γραμματεία εξέτασε και πάλι τις αναφορές αυτές και ας πούμε τις, ε, την ε, άσχημη αντιμετώπιση συμπεριφορά νεο, ε, νεογέννητων παιδιών σε ισπανικά νοσοκομεία κρίθηκαν παραδεκτές. Βέβαια υπάρχει και μια κάποια εξέταση, ανάλυση από πλευράς της δικαστικής ε, αρχής. Γι' αυτό ακριβώς διακόπτουμε την εξέταση αυτής της αναφοράς. Περιμένουμε την δικαστική απόφαση. Επίσης ε, είχαμε ζητήσει και σε άλλα θέματα από, για το θέμα της Λοβακίας ε, ορισμένες διευκρινήσεις ε, και αποφασίσαμε να δούμε και πάλι από την αρχή τα πράγματα σε μια συνάντηση όμως που θα συμμετάσχουν μόνο μέλη της Επιτροπής και εκπρόσωποι των αρχών των διαφερμένων χωρών χωρίς ε, δημόσια συμμετοχή. Και επίσης η αποστολή στη Δανία και αυτά που συζητήσαμε σε προηγούμενη συνάντηση για τα δικαιώματα ανηλίκων στην Δανία και θα ε, έχουμε το σχετικό πρόγραμμα σε λίγες μέρες. Επίσης, στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας θα έχουμε τις αναφορές που έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων στην Ιταλία, γιατί μετά από την εργασία παλαιότερων μηνών λάβαμε και μία λεπτομερή έκθεση από πλευράς ε, την αρχών για τον ανταγωνισμό των Ιταλικών ακριβώς που προσφέρει απαντήσεις στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην Επιτροπή μας. Α λοιπόν θα δοθεί συνέχεια στην εξέταση των ετοιμάτων των πολιτών. Και ακόμα το Προεδρείο εδώ έχει ζητήσει μέχρι την Πέμπτη το πολύ να έχουμε τις παρατηρήσεις για αυτό το συνοπτικό κείμενο των εργασιών της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών για το Way Days ε, που οργανώθηκαν το μήνα που μας πέρασε και ασχοληθήκαμε με διάφορα σημεία σημαντικά για την Επιτροπή μας. Οι συντονιστές δεν εξέτασαν άλλα σημεία. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις τότε μπορούμε να εγκρίνουμε όπως σας ε, εξήγησα μόλις τα συμπεράσματα των συντονιστών. Δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση, αλλά λοιπόν... Α, μισό λεπτό. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συμφωνία που επετεύχθη στην ε, συνάντηση των συντονιστών και για τις αναφορές Ισπανών πολιτών που έχουν να κάνουν με την απαγωγή νεογέννητων ε, στην Ισπανία από το 1940 μέχρι το 1990. Και επίσης να πω ότι καλό θα ήταν ήρεμα να εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε αναφορά λόγω της φύσης τους γιατί βλέπουμε ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε ξεχωριστά στοιχεία και εκεί, εκεί που θα, θα αρνηθούν να μας προσφέρουν πληροφορίες θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών να μην ε, το αναβάλουμε επαόριστον και εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι εκεί που ασχολείται η δικαιοσύνη με τις περιπτώσεις αυτές να περιμένουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων όπου πρόκειται όμως για περιπτώσεις που αρνούνται να μας δώσουν πληροφορίες, τότε θα έπρεπε εμείς να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις αναφορές αυτές. Αυτά λοιπόν. Α, λοιπόν κάθε περίπτωση ξεχωριστά, κάθε αναφορά να την εξετάζουμε ξεχωριστά. Κατά περίπτωση. Εντάξει, λέει πρόεδρος, συνάδελφε, θα προχωρήσουμε όπως ε, μας συμβολεύσατε. Τώρα για το 2011-92 σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο σαν εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τις δύο πρώτες συζητήσεις που κάναμε, έχω καταθέσει εγκαίρως ελπίζω, ελπίζω να έχετε δει, τις τροπολογίες Πολλές από αυτές τις τροπολογίες έχουν προκύψει από τις δικές σας παρατηρήσεις. Ορισμένες είναι με δική μου πρωτοβουλία. Όλες όμως ε, προσπαθούν και αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Επειδή πρέπει να είμαι σύντομος όπως με ειδοποίησαν και επειδή είναι η πρώτη κουβέντα, θα αναφερθώ σύντομα στις πιο βασικές από αυτές τις τροπολογίες. Και μάλιστα με τη μορφή κατηγοριών, όχι αναλυτικά. Πρώτον, υπάρχουν 7 τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται και προσπαθούν να κατοχυρώσουν τις ρυθμίσεις της συνθήκης του άορχους. Δηλαδή τη συμμετοχή και ενημέρωση του κοινού σε όλη τη διαδικασία αυτή που συζητάμε. Αυτή είναι μια κατηγορία τροπολογιών. Δεύτερη κατηγορία τροπολογιών είναι δύο τροπολογίες που αναφέρονται στην διασυνοριακή ρήπανση Υπήρξε παρατήρηση από αρκετού συναδέλφου, γι' αυτό είπα ότι πολλά από αυτά είναι από τι δικέ σα παρατηρήσει και είναι σύμφωνα με τη συνθήκη του ΕΣΠΟ, ούτω ώστε να καλύπτουν τα μεγάλα έργα που ενδεχομένω έχουν διασυνοριακέ δυσμενεί επιπτώσει στο περιβάλλον. Και είναι σωστό. Δύο τροπολογίε εκεί. Τρίτη. Αρκετοί συνάδελφοι, σχεδόν η πλειοψηφία από τι προηγούμενε συζητήσει, είχαν αναφερθεί με ένα σκεπτικισμό όσο αφορά το αν μπορούμε να εξαιρέσουμε την περίπτωση έργων έκτακτης ανάγκης. Το μελέτησα το θέμα και όπως τα είδατε στην τροπολογία διατηρώ αυτή την εξαίρεση άμεσης ανάγκης βάζοντας ορισμένους αυστερότερους κατά τη γνώμη μου όρους ούτως ώστε να περιφρουρήσουμε από πιθανές καταχρηστικές αξιοποίησεις αυτής της ρήτρα, αυτής της εξαίρεσης. Σημειώνω με αστερίσκο ότι έχω υποβάλει σχετική ερώτηση στην Κομισιόν για να δούμε τελικά όλο αυτό, όλο αυτό το διάστημα ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πανευρωπαϊκά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις υπήρξε εξαίρεση από την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξαίρεση από την προηγούμενη οδηγία. Σημείο τέταρτο, επιμένω, το βλέπετε και στην τροπολογία, να διαγραφεί η περίπτωση που αναφέρεται στο ότι εξαιρούνται έργα που, που λύνονται, ρυθμίζονται με ειδική εθνική νομοθετική πράξη. Την, ε, τους λόγους τους έχω εξηγήσει και στις προηγούμενες τοποθετήσεις και επιμένω αν θέλετε και για την ομοιόμορφη ε, ε, αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Σημείο 5 υπάρχουν οι τροπολογίες που προσθέτω για να βάλουμε τους έξι νέους ορισμούς που αφορούν τη βιοπικιλότητα, την επανόρθωση, τους ειδικού εμπειρογνώμενες άρτιους κτλ, την ανεξαρτησία τους, τις κυρώσεις και τις ποινές. Σημείο 7. Μια ομάδα τροπολογιών αναφέρεται σε μια προσπάθεια που γίνεται να αποσαφινιστεί ποιος αποφασίζει και ποιος πρέπει να έχει ε, να δει ότι έχουν ε, γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων και πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η ουδετερότητα και η αμεροληψία. Σημείο 7. Θεωρώ ότι είναι θετική η προσθήκη για την παρακολούθηση. Υπάρχει μια κατηγορία τροπολογιών που και εκεί προστίθεται παρατηρήσεις και επισημάνσεις όσο αφορά το κοινό και την ενημέρωση του κοινού και τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται κατά την πορεία εκτέλεση των έργων από τον κύριο ε, του έργου, από τον ε, εκτελεστή. Τέλος, σημείο 8 και τελευταίο είπα ότι θα είμαι σύντομος, στα παραρτήματα που ακολουθούν την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας έχω υποβάλει ορισμένες τροπολογίες για να συμπεριληφθούν μεταξύ των οποίων αναφέρω για την υπόθεση της εξόριξης φυσικού αερίου και σχιστολιωδικού πετρελαίου Κυρία Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω, όπως είπα, εν συντομία και περιμένω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστώ. Ο κύριος Τανόνι είναι μαζί μας. Είναι εισηγητής από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ και τον κύριο Χουντή για τις ε, προτινόμενες τροπολογίες του. Δεν μπορούμε να διατρέξουμε κάθε μία τροπολογία, οπότε θα τις ομαδοποιήσω σε τρεις κατηγορίες. Αυτές που καλωσορίζουμε και σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν τα θέματα εποπτείας και οι διορθωτικές δράσεις, καθώς επίσης και η βελτίωση των παραρτημάτων. Επίσης η ενσωμάτωση του, του συμβάσεων ΕΣΠΟ και όρχους, στο βαθμό που βεβαίως μπορούμε να ορίσουμε περισσότερο τις απαιτήσει για αυτές τις δύο συμβάσεις, παρόλο που είναι τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, οπότε δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Και σε σχέση με την διασυνοριακή, τις διασυνοριακές επιπτώσεις που έχουν κάποιο από αυτά τα project, συμφωνούμε. Επίσης συμφωνούμε με, την, με τον επίγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με την υποβολή των εκθέσεων. Ο κ. Κοντούς έχει, ε, έχει δεχθεί να παραμείνει η πρόταση ως έχει στο σημείο αυτό. Περνάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία, όπου επί της αρχής συμφωνούμε, αλλά θα θέλαμε να μελετηθεί λίγο περισσότερο το πράγμα και να διευκρινιστεί. Εδώ μιλώ για τα εκτιμώντας, τις αιτιολογικές σκέψεις. Δεν θα θέλαμε να επαναλαμβάνονται αιτιολογικές σκέψεις που ήδη υπάρχουν στην ε, κωδικοποιημένη οδηγία που τροποποιείται από την πρότασή μας. Νομίζω ότι θα υπάρξει έτσι επικάλυψη με ιδεολογικές ε, σκέψεις που ήδη υπάρχουν. Μόνο αυτές που χρειάζονται για να, να αιτιολογηθούν οι προτάσεις που υπάρχουν, ή διατάξεις στην, τροποποιημένη, στην τροποποιητική πρόταση μάλλον. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα εκτιμώντας. Τώρα για τους ορισμούς. Ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για ορισμούς και η δική μας ανησυχία είναι ότι ε, δίνουμε ορισμούς για κάποια σημεία ενώ δεν δίνονται ορισμοί για κάποια άλλα. Ας πούμε, ε, όπου υπάρχει ανάγκη να, παράχει, να παρέχεται ορισμός, καλό θα ήταν αυτό να γίνεται στο άρθρο. Τώρα, πάμε στην τρίτη ομάδα, όπου επί της αρχής είμαστε αρνητικοί με τα όσα προτείνονται, με τις προτινόμενες τροπολογίες δηλαδή. Μιλούμε για τις κυρώσεις και τις ποινές, κυρίως αυτές που συνδέονται με τις δραστηριότητες των πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων. Συμφωνούμε ότι αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και γι' αυτό μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία που αναφέρεται στην ανεξαρτησία και στην ε, αντικειμενικότητα των ε, εμπειρογνωμόνων αυτών ε, των διαπιστευμένων, αλλά το να συνδέονται οι δραστηριότητε του με κυρώσει και ποινέ, μάλλον ξεπερνά το πεδίο εφαρμογή και τη νομική βάση αυτή τη πρόταση. Μια που στην συνθήκη της Λισαβόνα υπάρχει συγκεκριμένη νομική βάση για τις κυρώσεις και τις ποινέ που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε τούτη την πρόταση και δεύτερον υπάρχει και ε, μια οδηγία για την περιβαλλοντική εγκληματικότητα που το ξέρετε, την ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό. Θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να εφαρμοστεί. Ε, η άλλη, ε, η άλλη ομάδα τροπολογιών είναι, αφορά άρθρα που δεν καλύπτονται από την πρόταση αναθεώρησής μας. Άρθρα δηλαδή που δεν έχουμε πειράξει και που δεν έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα στην ομάδα εργασία στο Συμβούλιο. Παράδειγμα, πρόσβαση στη δικαιοσύνη και οι σχετικές διατάξεις, άρθρο 11 δηλαδή, και το συστολιστικό αέριο. Βεβαίω, υπό το φω των συζητήσεων που θα γίνουν στο μέλλον, ε, προφανώ θα υπάρξει κάποιο είδου συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, που θα δούνε πώς θα μπορούσε αυτό να συμπεριληφθεί. Αλλά σε τούτη τη φάση που είμαστε δεν μπορούμε να δεχτούμε τη θέση που υπάρχει ως προς το θέμα αυτό. Και σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τα project που μπορούν να ε, επιτραπούν μέσω εθνικής νομοθεσίας, μέσω εθνική νομοθετική διαδικασία, που δεν είναι η οποιαδήποτε νομοθετική διαδικασία, αλλά που πρέπει να έχει τύχει και κάποια αξιολόγηση, δηλαδή τροπολογία 17. Δεν είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτή η δυνατότητα ήδη προβλέπεται στη Σύμβαση Όρχους και γι' αυτό ως τέτοια είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Επομένως, ε, τροποποιούμε μία διάταξη η οποία είναι κομμάτι του κεκτημένου. Και επιπλέον, η πράξη δείχνει ότι αυτή η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και η εμπειρία επίσης δείχνει ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε πρόβλημα εφαρμογής σε σχέση με τούτη την οδηγία. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Μπέλιε. Ναι, η κυρία Μπέλια, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ εισηγητή για την εργασία του, για την οδηγία αυτή, για τις επιπτώσεις ορισμένων σχεδίων ιδιωτικών και δημοσίων στο περιβάλλον και για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εγώ είμαι εισηγήτρια ξεκινήσαμε την εργασία μας με τον κύριο Ζανόνη θα ήθελα να προβώ σε ορισμένε παρατηρήσει και αν δεν υπήρχαν προβλήματα τότε δεν θα μιλούσαμε καθόλου για αναθεώρηση για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί καλύτερα από τα κράτη-μέλη στο επικράτεια τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω την εργασία στην Επιτροπή περιβάλλοντο. Ποια ήταν αυτή. Ε, συνένεση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η αναθεώρηση από την Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζουμε ότι θα καλύψει τα κενά της οδηγίας αυτής τα κενά εφαρμογής και το πεδίο εφαρμογής. Επίσης, οι ιδιαίτερες σπουδές ε, βελτιώσεις για τη ρύθμιση επίσης και την ανιχνεύση και ε, ε, για όλα αυτά τα σχέδια, να δούμε καλύτερα τα πράγματα για εναλλακτικέ λύσεις, για να δούμε ε, κατά ποιο τρόπο το δημόσιο θα συμμετέχει, επίσης προσφυγή στη δικαιοσύνη ενδεχόμενα. Και αυτή η εργασία απέναντι στον εισηγητή νομίζουμε ότι προχώρησε καλά και θα η εργασία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν ιδιαίτερα θετική και προσφέρεται μια νομιμότητα έτσι που βασίζεται σε αρκετές εμπειρίες και εδώ στην Επιτροπή αναφορώ γιατί πόσα πολλά για αεροδρόμια, για οδικά θέματα κλπ. μας κινητοποίησαν στην σχετική εκτίμηση επειδή δεν ε, σεβόταν τις προδιαγραφές. Ε, εδώ θα ήθελα να καταλήξω, να ολοκληρώσω, να πω ότι εξ των οικολόγων ε, παρακαλώ προσέξτε την 48 τροπολογία που οπωσδήποτε θα πρέπει να υποστηριχθεί από τα μέλη της Επιτροπής μας. αντά αφορά τις μη συμβατικές μεθόδους σχιστικού αερίου και επίσης ε, αεροποίηση κάρβουνου, παρόμοιες μεθόδους. Ε, εδώ απευθύνθηκαν πολλοί πολίτες ε, γιατί πραγματικά τους απασχολεί ο κίνδυνος από τις νέες αυτές μεθόδους εξόριξης. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσουν το περιβάλλον αλλά ίσως πρέπει να δημιουργηθούν ανησυχίε. Άρα λοιπόν στο παρατημά τη οδηγία να μπουν αυτά τα πράγματα για να δούμε ότι πρώτα απ' όλα υπήρχε μια σωστή εκτίμηση και ότι λήφθηκαν σοβαρά υπόψη πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βάλιαν. Yes. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χουντή για τις τροπολογίες του και να κάνω κάποια σχόλια για τότε την νομοθετική πρόταση. Όπω πολλέ από τις αξιολογήσει επιπτώσεων που ζητούμε να γίνουν, ε, αυτή η οδηγία νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσει σε τρεις διαφορετικές απαιτήσει. Καταρχάς, να εξασφαλίσει ότι το περιβάλλον θα προστατεύεται, όπου και όποτε υπάρχει νέο project. Δεύτερον, να ενημερώσει το κοινό, που το αφορά βεβαίως, και να μειώσει την γραφειοκρατία για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, καλωσορίζω την πρόταση τη Κομισιόν για μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινή νόμη στις όλες διαδικασίε Παρ' όλα αυτά. Η υπεποίθηση ότι η γραφειοκρατία είναι το κλειδί ώστε να, είναι, να δείξουν λογοδοσία οι εταιρείε δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί όλοι οι αναφέροντε που έχουμε δει σε τούτη την Επιτροπή έχουν δείξει ότι η τεκμηρίωση και οι εκθέσει δεν εξασφαλίζουν την σωστή εφαρμογή. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι υποχρεώσεις ε, για τους ε, ε, εκτελεστές για την παροχή πληροφοριών είναι δυσανάλογες. Ε, η υποχρέωση να, παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν ε, ληφθεί είναι νομίζω πολύ προβληματική. Αυτό σημαίνει ότι ε, ο έλεγχος ξεπερνά τα όσα προβλέπονται ή τα όσα σημαίνουν, ε, σημαίνει μία αξιολόγηση επιπτώσεων, δηλαδή η τα οσα σημαινουν σημαινει μια αξιολογηση επιπτωσεων δηλαδη η αναλυση για τα μελλοντικά project. Μία σαφής παρουσίαση σε τούτη τη φάση κάποιων άλλων μέτρων νομίζω λοιπόν ότι είναι πρόορη. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το θέμα του ETS. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε επικάλυψη νομοθετικών κειμένων. Δεν είναι απαραίτητο να, να λαμβάνουμε υπόψη και τις εκπομπές που καλύπτονται από το ETS ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, σε τούτο το κείμενο. Και επίση υπάρχει υποχρέωση οι developers να παρουσιάσουν και εναλλακτικέ στα project σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική του έκθεση. Αλλά αυτό σημαίνει επιπλέον διοικητικό βάρο. Οπότε του ζητούμε ουσιαστικά, ζητούμε από μια εταιρεία να βρει εναλλακτικέ, πιθανέ εναλλακτικέ με το χαμηλότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον αλλά αυτά τα προγράμματα δεν υπόκεινται ούτε σε EIA, ούτε είναι σε φάση προγραμματισμού ή σχεδιασμού. Και αυτό κοστίζει και χρόνο και χρήμα. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, θα πρέπει να δείξουμε ε, ευελιξία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να συμφωνήσω με τον κύριο Χουντή σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στην τροπολογία που έχει υποβάλει για τις πιο αυστηρούς κανόνες για τους, επιπλέον, ε, τις επιπλέον κυρώσεις, τα πρόστιμα, τις παρεκκλήσεις λόγω της εθνικής νομοθεσίας. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερέστερα τα σημεία αυτά για να μπορέσουμε να βρούμε μια ε, ισόρροπη προσέγγιση. Να δούμε τι, έχει, τι περιλαμβάνει η νομοθεσία που έχουμε και πρέπει να πω ότι τα, επιπλέον ποινέ και τα πρόστιμα και η γραφειοκρατία ποτέ δεν καταφέρουν το στόχο του. σω να πρέπει να ζητήσουμε απόδειξη συμμόρφωση, πρέπει να δείξουμε μια ευελιξία παρόλα αυτά για να καλύψουμε ε, τα αιτήματα των εταιριών και βεβαίω ε, θα περιμένουμε χαρά να συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Βαλιάν, ο κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι Είμαι πολύ χαρούμενος με την πρόταση αυτή του αγαπημένου συναδέλφου, του κυρίου Χουντή, γιατί η δική του η συμβολή δείχνει καταρχάς πόσο σημαντικό είναι για την Επιτροπή Αναφορών το να ασχοληθεί με τις ανησυχίες των πολιτών. Έχουμε δει τόσες πολλές αναφορές σε, σε αυτή την χρονική φάση που δείχνει ότι πάντα υπάρχουν ε, γέφυρες σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι σε μερικά, σε όλα τα κράτη-μέλη, από τα πιο ανεπτυγμένα στα λιγότερο ανεπτυγμένα ή στα, στα, μέλη που ε, πρόσφατα, ή τέλο πάντων τόσο πρόσφατα, αλλά μετά το 2004 μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Δεύτερον, θα πρέπει να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι, Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκές κοινότητες. Αυτό θα πρέπει να το δούμε άμεσα. Και είναι σημαντικό να δούμε το πρόβλημα της ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων αντικτύπου που νομίζω ότι το έχει παρουσιάσει πολύ καλά ο κύριος Καλώς Καλωσορίζω λοιπόν το σημείο αυτό. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι ενώ έχουμε την, ε, τις συμβάσεις όρχους και ΕΣΠΟ και εφαρμόζονται, θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στη δική μου εμπειρία για τη Ρουμανία και την Ουγγαρία που ε, συζητούν ένα κοινό ε, project το οποίο δεν το διαχειριστήκε σωστά η Ρουμανία, δεν ήθελε να δώσει στην ουγγρική πλευρά τις απαραίτητες πληροφορίες και στο τέλος δεν τους ενδιέφερε κιόλα να εμπλακούν οι Ούγγροι σε αυτό, το, ε, σε αυτό το project. Οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Η, η ολοενημέρωση πρέπει να βελτιωθεί. Επίσης, πρέπει να δούμε τις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες η στρατηγική αξιολόγηση δικτύπου για το περιβάλλον θα εφαρμόζεται σωστά. Γιατί ε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα, και από ό,τι μου έχει πει και πρόσωπο από την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο, αυτή η τακτική τη σαλαμοποίηση υπάρχει, αλλά δεν, δεν είναι ικανοποιητική. Μπορεί να εφαρμόζεται παντού στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ικανοποιητική όταν χρειάζεται στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση αντικτύπου. Όταν θέλουμε να λαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία υπόψη, τότε δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος πέραν της στρατηγικής αξιολόγησης, περιβαλλοντικής αξιολόγησης αντικτύπου. Και επίσης, στις δύο με προσκάλεσαν να μιλήσω για την ε, Ευρωπαϊκή Γεωλογική Έρευνα εκπροσωπώντας τα 28 κράτη-μέλη, τα 27 συν 1, εν πάση περιπτώσει, σύντομα θα μπει και η Κροατία. Και μου είπανε ότι όταν, όταν συζητούμε το νέο κείμενο του κανονισμού, το νέο σχέδιο, τόσο τόσοι πολλοί ε, ε, τόσο πολλοί ε, φορεί εκτό από την Ευρωπαϊκή Γεωλογική Έρευνα. Και καλούν το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη τη γεωλογική διάσταση τη περιβαλλοντική αξιολόγηση αντικτύπου. Γιατί είναι προφανέ ότι σε σχέδια που έχουν σχέση με τον τομέα τη ενέργεια, με, την, το, με τον κλαδό τη εξόριξη ή με τι πρώτε ύλε, είναι θεμελιώδες, είναι ουσιώδες να διερευνήσουμε και, τον αντίκτυπο στα γεωλογικά στοιχεία των μελλοντικών project. Και αυτό πραγματικά είναι, ε, μιλούμε για ανθρώπους, και μια κοινότητα επιστημόνων που είναι αφοσιωμένοι σε αυτό και θα πρέπει η φωνή τους να μπορεί να ακουστεί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δικό μας καθήκον ως Κοινοβούλιο να ε, καταστήσουμε ε, δυνατή την δική τους τη φωνή. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Ζανόκα. Στο επόμενο σημείο, Πρόεδρε, δεν ήθελα το λόγο για, το, για τούτο. Κύριε Χουντή, θέλετε το λόγο. Conclude. Πολύ σύντομα, όπως και τα αρχικά σχόλια που έκανα, ε, θέλω να ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις που έγιναν. Ε, η συνόψιση έγκυται στο εξής, πάλι κωδικοποιημένα. Σημείο πρώτο. Θέλω να θυμίσω ότι δουλεύουμε πάνω σε μία οδηγία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είναι ένα πολύ κρίσιμο εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και που θα πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Σημείο δεύτερο. Η τροποποίηση που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Κομισιόν αλλά και που προτείνουμε και εμείς πρέπει να την κάνει πιο αποτελεσματική την εφαρμογή βεβαίως και την ίδια την οδηγία. Θέλω σημείο τρία. Η Επιτροπή και εμείς από τη μια πλευρά διαπιστώσαμε ότι λόγω ελλειπούς εφαρμογής, όχι εναρμόνισης κτλ. είχαμε προβλήματα. Και εδώ χιλιάδες οι αναφορές όλα αυτά τα χρόνια στην Επιτροπή Αναφορών για αυτό το θέμα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έκρυψα από την αρχική τοποθέτηση του ζητήματος ότι η τροποποίηση της οδηγίας σε τούτους τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, καιρούς κρίσης και ύφεσης, όπου η ανάγκη για αναπτυξιακές δραστηριότητες πολλές φορές τίθενται ως πρώτη προτεραιότητα για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της ύφεσης και το περιβάλλον πάει ως δεύτερη προτεραιότητα, αυτό είναι ένα σημείο που κατά τη γνώμη μου πρέπει να, η Επιτροπή μας να το προσέξει πάρα πολύ. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, έχω άμεση εμπειρία, δεν σας κουράζω περισσότερο. Σημείο πέμπτο, κατόπιν και αυτών των σκέψεων, σχετικά με την αναφορά του εκπροσώπου της Κομισιόν, τον ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, αυτά που καλωσορίζει έχει καλώς, νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, έχουμε κάνει και μια σχετική συζήτηση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, εφόσον έχουμε να, ασχοληθούμε με τροποποίηση οδηγίας δεν περιοριζόμαστε να καταθέσουμε τροπολογίες μόνο σε ό,τι έχει καταθέσει η Κομισιόν. Μπορούμε να καταθέσουμε και δικές μας τροπολογίες και σε άρθρα που δεν θίγει η πρόταση της Κομισιόν. Άλλωστε αυτή είναι η ενεργητική νομοθετική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ειδικά της Επιτροπής μας Αναφορών και αυτό το δικαίωμα, αυτού του δικαιώματος έκανα χρήση και σε ορισμένα πράγματα πρότεινα κάτι που δεν το έχει προτείνει η Κομισιόν και νομίζω ότι είναι σημαντικό όσον αφορά τη θεσμική ισορροπία μας σε σχέση με την νομοθετική διαδικασία σε, όλη την, ε, ε, ε, σε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δύο πράγματα πιο συγκεκριμένα σχετικά με τον επίγοντα χαρακτήρα και την εξαίρεση που διατηρώ ξαναλέω έτσι είναι τα πράγματα την κάνουμε πιο αυστηρή έχω ακόμα επιφυλάξεις εφόσον δούμε και τα στοιχεία όλο αυτό το διάστημα που έγιναν εξαιρέσεις σε τέτοιες περιπτώσεις αν εμπεδώνεται η ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες εξαιρέσεις όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Η πρότασή μου όμως είναι σαφής να την κρατήσουμε και να έχουμε διαφορετικά πράγματα. Τώρα για τις κυρώσεις και τις ποινές, τώρα ένα σχολιάκι έτσι γενικότερο. Εφόσον πια ε, μέσα στο γενικό κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Έχουμε περάσει σε ποινές και κυρώσεις ολόκληρων κρατών ε, όταν κατά τους δείκτες και δεν κρατάνε κάποια πράγματα γιατί φοβόμαστε να είμαστε πιο αυστηροί εκεί. Όταν δηλαδή οι εμπειρογνώμενες δεν τα έχουν κάνει καλά τα πράγματα. Το σχήμα νομίζω το καταλάβαμε. Έτσι αφού περάσαμε σε μια κυρωτική διαδικασία και ποινή, το αξιοποιώ και εγώ, <laughs> να σα το πω έτσι απλά, να είμαστε αυστηροί και μάλιστα σε περιπτώσει που έχουμε επιδράσει άμεσα στο περιβάλλον και από αφορά πρόσωπα, εταιρείε κτλ. κτλ. Λοιπόν, και το τελευταίο για την ειδική, ε, να μην εξαιρούνται αυτά που κανονίζονται με ειδικέ εθνικέ νομοθετικέ πράξει. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε επόμενη συζήτηση μπορώ να σας πω τι γίνεται σήμερα, κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα, όπου γίνονται διάφορα σημεία και τέρατα σε βάρος του περιβάλλοντος στο όνομα ότι αυτό το έργο, αυτή η δραστηριότητα έχει καθοριστεί για ειδική <laughs> νομοθετική δραστηριότητα. Αυτό είναι και ο φόβο μου, αγαπητοί συνάδελφοι, και θέλω να σα το πω. Στο όνομα γενικότερων αναγκών. Κατά τα άλλα, οι παρατηρήσει είναι πολύ χρήσιμε. Όπω ξεκίνησα παίρνοντα υπόψη και τι παρατηρήσει των συναδέλφων, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να κάνει μια συλλογική αποτελεσματική δουλειά υπερασπιζόμενη και το κύρος της ιδιαίτερα σε θέματα που έχουμε τόσες και τόσες αναφορές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Χουντή, σας ευχαριστούμε. Αυτό το προσχέδιο του κυρίου Χουντή θα εξεταστεί στις 24 Απριλίου και προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 7 Μαΐου 27-28 Μαΐου η εξέταση τροπολογιών... και 19 Ιουνίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Έτσι, καμία άλλη ανακοίνωση, άρα λοιπόν μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μετά από τις αλλαγές μας, σήμερα το πρωί στην ημερήσια διάταξη, θα ασχοληθούμε με το σημείο 14 τις τρεις αναφορές του σημείου 14. Είναι του ε, Τσέπμα στην ε, Notre Dame de Land την κατασκευή αερολιμένα Επίσης ε, για το ίδιο θέμα άλλη μια αναφορά και από τον Μπρουν Σβέντι εξ ονόματος της France Natural Environment για το ίδιο σχέδιο κατασκευής. Τέσσερις έχουν υπογράψει, τέσσερις είναι οι αναφέροντες και θα μας εκθέσουν το θέμα τους. Παρακαλώ όμως να σεβαστούν το χρόνο μιλίας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα την όλη συζήτηση. Έτσι, το πολύ λοιπόν πέντε λεπτά ο καθένας. François Κυρίες, κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, σήμερα είμαστε μπροστά εξ ονόματι 40.000 πολιτών, 1.200 ερωτών εκπροσώπων και εκ μέρους πολλών γεωργών και από μέρους συνδικάτων. Εμείς αμφισβητούμε την ανάγκη να υπάρξει το νέο αεροδρόμιο κοντά στην Άντι και ο τόπος τον οποίο έχει επιλεχθεί. Αυτός ο τόπος στην notre Ντάμστιλαντ, στη ε, έχει επιλεγεί πριν από 50 χρόνια. 98%, ε, χρόνια, 98 του εδάφους είναι υδρόφιλες περιοχές, ε, στις περιοχές του Λουάρ και του Βιλέν και έχουμε μια μεγάλη παραγωγή προϊόντων γάλακτος η οποία κινδυνεύει από τη δημιουργία αυτού του σχεδίου. Είμαι Γιώργος και μπορώ να δώσω εδώ την απόψη μου σε σχέση με αυτή τη μεγάλη υδρόφιλη περιοχή. Εμείς κάνουμε, παράγουμε γάλα, στα πλαίσια πάντα συμβατά με τη νέα ΚΑΠ. Όλοι οι οργανισμοί των γεωργών καταγγέλνουν αυτή την ε, προσπάθεια και τον τρόπο τον οποίο καταστρατηγείται η περιοχή μας. Αυτό θα οδηγήσει στην ε, εξαφάνιση 15 μονάδων παραγωγή και 500 ε, θέσεων εργασία. κάτι για το οποίο δεν μιλάει κανεί. Επίση, έχουμε παρουσία στρατιωτική τις τελευταίου 6 μήνε. ε, δύσκολες συνθήκες και προσπάθειες να μας αναγκάσουν να φύγουμε. Οι δυσκολίες είναι καθημερινές, συνεχείς, ε, για να μας αναγκάσουν να φύγουμε. Η αντίσταση όμως είναι μεγάλη. Εμείς θέλουμε να μείνουμε επιτόπου, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τη γη, να έχουμε τα ζώα μας, και να εμποδίσουμε την καταστροφή αυτή τη περιοχή. Η γεωργία έχει μέλλον και μπορεί να δημιουργήσει θέσει εργασία. Αλλά φυσικά πρέπει να την αφήσουν στην ησυχία τη. Για μα αυτό το σχέδιο αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο για πολλού τρόπου. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο για το νερό, τι υδρόφιλε περιοχέ, του κατοίκου και τα διάφορα ε, είδη ζών. Ο διάλογο στη Γαλλία γίνεται σε σχέση με το θέμα που έχει φορά το, τα ύδατα ε, άρχισε μόλις το 2012 ενώ έχουμε δημόσιο διάλογο ήδη από το 2003 και από το 2008. Επιμένει η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση στη θέση της που έχει να κάνει με τα δικαιώματα στη γη και αυτά ξεκινούν από το 1973. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι αμερόληπτο και ποτέ δεν ε, έκανε εναλλακτικέ προτάσεις για και για να μποράσει να προχωρήσει αυτά τα σχέδια τα αρνητικά προσπαθεί να παρακάμψει τις ε, θεμελιώδεις αρχές για τα ύδατα. Επίσης έχουμε να κάνουμε με έναν τρόπο οικονομικής διαχείρισης όπου προσπαθεί με τον ένα ή αλφα τρόπο άμεσες επιδοτήσεις και άλλους να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα. Έχει γίνει μια έρευνα από γραφείο Ολλανδικό εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας δείχνουν ότι έγινε μια εκτίμηση όσον αφορά το όφελο κέρδο στο αρχικό σχέδιο. Ο νέος, το νέο αεροδρόμιο που μας παρουσιάζεται σήμερα ε, δεν, ε, δεν έχει σχέση να κάνει με τίποτα με αυτό που ήταν το αρχικό σχέδιο. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει ε, ε, ανάγκες, περισσότερες ανάγκες από το παλαιότερο. Αναφέρεται ο αριθμός των 4,5 εκατομμυρίων επιβατών, ενώ το, το, το, τωρινό καλύπτει 4 εκατομμύρια ε, επίσης προβλέπουν 10.000 θέσεων παρκινγκ οριζόντια, το οποίο ε, θα χαλάσει πολύ γη θα λέγαμε. Το σημερινό αεροδρόμιο είναι ήδη διεθνές και μπορεί κανείς να το βελτιώσει, μπορεί να κανείς να το μεγαλώσει για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες. Μπορεί επίσης να εξυπηρετηθεί από το, τα, τα τρένα ή τα τραμ. Ε, όλα είναι βελτιώσιμα. Και, και σήμερα βλέπουμε ότι γίνονται ενέργειες ε, οι οποίες δεν χρειάζονται να γίνουν για να μπορέσει κανείς να βελτιώσει τις υπάρχουσες ε, ε, εγκαταστάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι άμεσο το πρόβλημα διότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μια μη αναστρέψη κατάσταση. Φαίνεται ότι θα αργήσουν εργασίες τις επόμενες μέρες. Συνεχίζονται οι να καταστρέφονται κτίρια και έχουμε και τις αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνονται κάτω από στρατιωτική προστασία. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε ένα αγώνα ε, ε, ε, με το χρόνο και εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό, πρέπει να γίνουν σεβαστές οι οδηγίες της Ευρώπης. Δεν πρέπει να χαθεί ε, καλλιεργήσιμη γη. Επίσης χρειάζεται να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα και γι' αυτό το λόγο κάνουμε μια έκκληση σας να έρθετε επί τόπου να δείτε το υπάρχον αεροδρόμιο και αυτό το οποίο προτείνεται στην Notre Dame της Λάντα. Θα καταλάβετε δηλαδή γιατί πρέπει να κινητοποιηθούμε για να αποφύγουμε το μη αναστρέψιμο. Η αντίσταση που υπάρχει επί τόπου και παντού στη Γαλλία ε, μαρτυρεί την ανάγκη αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε λέει και η πρόεδρος. Ο κύριος Bon, Καλώς, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε κύριοι βουλευτές, κυρίες κύριοι και σε όλους τους άλλους. Σας ευχαριστώ που θεωρείτε ότι ε, ε, είναι αποδεκτή η, αναφορά μας από τον Σεπτέμβριο του 2012 έχουμε να κάνουμε αυτό το θέμα του αεροδρομίου στη Λάντ και οδήγησε αυτή η κατάσταση σε αυτή την αναφορά. Η Δυτική Γαλλία, δεν βλέπω να, ε, τις διαφάνειες, για να καταλάβει κανείς θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα. Να λειτουργήσουν λειτουργήσουν οι διαφάνειες λοιπόν. Ça marche, Marc Non Sabotage. Σαμποτάζ λέει ο μιλητής. Μας κάνει. Μπορούμε κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Euh. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη δεύτερη σελίδα, στην επόμενη μάλλον, εκεί. Βλέπετε τη Δυτική Γαλλία, μια ε, περιοχή με 8 εκατομμύρια κατοίκους που είναι, ε, θα λέγαμε, από, απόμακρη από τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Απ' την άλλη έχει ε, δυσκολίες με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και με το ΤΕΖΕΒΕ ακόμα στη Γαλλία. Ε, το σημερινό αεροδρόμιο ε, έχει μια αύξηση στην κινητικότητά της Εδώ πέρα όμως περιμένουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα ένα εκατομμύριο επιβάτης σε αυτό το αεροδρόμιο μέχρι το 2030. Ε, απ' την άλλη βλέπουμε ότι ο κόσμος ε, θα έχει μεγάλα προβλήματα με το θόρυβα. 40.000 άτομα εκτίθενται σε αυτό. Τα αεροπλάνα πετάνε πολύ χαμηλά και, και απάνω από μια περιοχή και λίμνη οι οποίες είναι στο προστατευόμενες. Υπάρχει ένα πρόβλημα δεν μπορούν να δημιουργηθούν οι προτινόμενες πίστες για το προσγείωση σύμφωνα με μελέτε που έχουν γίνει. Αλλά σε σχέση με αυτά που λένε, η μεταφορά του αεροδρομίου δεν θα οδηγήσει σε επιπτώσεις που αναφέρονται σε σχέση με τους γεωργούς. Υπάρχει το θέμα της ε, φιλικής ε, διαχείρισης. Όλο και πιο πολλοί νέοι ε, καλλιεργητές εγκαθίζονται στην περιοχή για την... το περιβάλλον. Μόνο ένα μικρό ποσοστό της επιφάνειας έχει χρησιμοποιηθεί και υπάρχει μια περίμετρο προστασίας των φυσικών χώρων και αυτό έχει εξασφαλιστεί. Έχει... Και σε σχέση με, αυτά το κράτος έχει δώσει σύμφωνη τη γνώμη, φαίνεται ότι προστατεύεται η φύση και σίγουρα θα εγγυάται την δημιουργία μιας επιτροπής επιστημονική η οποία θα διασφαλίσει το θέμα που έχει να κάνει με τα ύδατα. Γίνονται επίσης προσπάθειες να προβλεφθούν κάποιες ε, διαβολεύσεις ε, που είναι απαραίτητες για ένα σχέδιο αυτής της έκτασης. 41 εκατομμύρια διατίθεται για αυτό το θέμα. Είναι ένα παραδειγματικό θα λέγαμε σχέδιο όσον αφορά τις ψυχές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον γίνονται σεβαστές ε, όλες οι αρχές που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη έχει απορρίψει όλα τα αντίθετα επιχειρήματα. Το αεροδρόμιο ε, στα πλαίσια του νόμου ε, του 79 ε, διαγράφεται στα πλαίσια της διαχείρισης της επικράτειας της χώρας. έχει επαληθευθεί ε, το 2009 η μεταφορά αυτού του αεροδρομίου και αυτά στα πλαίσια της, οδηγίας, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων αεροδρομίων που θα ακολουθήσουν κάποιους περιορισμούς. Και ε, έχει εγκριθεί αυτό το αεροδρόμιο, αυτή η μεταφορά και σε μια οικονομική και κοινωνική συγκυρία αρνητική αυτό το σχέδιο είναι πολύ σημαντικό διότι θα δημιουργήσει ε, θέσεις εργασίας 4, ε, εκατομμύρια ώρες εργασίας σε μια περιοχή η οποία ε, έχει δύο ε, ε, βιομηχανίες που έχουν να κάνουν με την εργασία και άλλες. Επιπλέον, να σας πω και η μακροπρόθεσμα πώς θα λειτουργήσει αυτό. Διότι αυτό το σχέδιο έχει να κάνει με τις επόμενες δεκαετίες της Δυτικής Γαλλίας που θα δεχθεί 1,5 εκατομμύριο νέους κατοίκους μέχρι το 2040. Και είναι σημαντικό, φέρει χώρες σαν την Αυστρία, τη, τη Σουηδία, ε, ε, Τι γίνεται, πρέπει να κανείς να κλειστεί στον εαυτό σου, να υποχωρήσει. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ε, ε, παρεθοντολόγοι. Σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε κάποιες αρχές και με ένα ορθολογικό τρόπο να προχωρήσουμε αυτό το σχέδιο. Ένα αεροδρόμιο υψηλής ποιότητας όσον αφορά το περιβάλλον, σωστή κατανάλωση ενέργειας που θα είναι ε, στο 1 τρίτο από του σε σχέση με αυτό που καταναλώνει το υπάρχον αεροδρόμιο. Είμαστε πριν από τις εκλογές τις ευρωπαϊκές και οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούσαν μια ε, Ευρώπη η οποία να ε, μην οδηγείται σε κυρώσεις αλλά να προχωρεί προς τα μπράς. Και για να μπορέσει δηλαδή να είναι ελκυστικό ο χώρος, η περιοχή μας και να προχωρήσει, αυτό το σχέδιο αποτελεί μία προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. The floor to Mr. Bruno Genti. Ο κύριος Bruno Genti έχει το λόγο. Τελευταίος ομιλητής. C'est amusant parce qu'il faisait que tout à l'heure, il plus On va prendre le pouvoir. Ah, euh, Madame la Présidente. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την υποδοχή σα Μπρούνο Τζάντι από την Γαλλική Ομοσπονδία των Ανώσεων ε, προστασία ε, του περιβάλλοντο. και θα ήθελα να υποστηρίξω αυτή την αναφορά που υποβάλαμε μαζί με πέντε ακόμα ενώσεις ή τέσσερις μέλη του France Nature Environnement. 800.000 έχουμε που μας υποστηρίζουν αλλά και με διάφορες ε, ενώσεις επιτόπου. Εδώ για το σχέδιο για το αεροδρόμιο, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη ένα σχέδιο σε 200, 1200 κτάρια, κάπου που προστατεύεται, είναι φυσικός τόπος με υψηλής ποιότητας και περιοχή με υψηλή υγρασία στην περιοχή εκείνη και με βιοπικιλότητα η γαλλική κυβέρνηση τον έκανε, έκανε αυτή την αλλαγή πολιτικό στόχο αλλά ε, το σχέδιο είναι κατά του στόχου της κυβέρνησης του παλιότερου αυτού. Εμείς γιατί τα προτείνουμε αυτά. Υπάρχουν νομικά θέματα που προκύπτουν από τα διάφορα κοινωνικά και ο συνάδελφος ε, νομικός θα μας πει πως έχουν τα διάφορα προβλήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή αυτή οδηγία. Απλά και μόνο να κληρώσω με τα εξή λόγια, ότι είναι κατεπήγον το θέμα, αλλά έχουμε το χρόνο να αντιδράσουμε. Εδώ είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, είμαστε στον οίκο του Ευρωπαίου πολίτη. Παρακαλώ ελάτε, ελάτε να δείτε το αεροδρόμιο που υπάρχει ήδη και το Δόπο που σχεδιάζεται το νέο αεροδρόμιο. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Έξι σημεία που δεν σέβονται το δίκαιο το κοινοτικό. Δύο σχετικά με τις οδηγίες για τα προγράμματα, γιατί το σύνολο αυτών των στοιχείων θα πρέπει να ένα πρόγραμμα σύμφωνα με την οδηγία του 2001 και να βλέπουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι επιπτώσεις αυτές, οι εκτιμήσεις αυτές και με τη συμμετοχή ε, που θα έπρεπε να υπάρχει χωρίστηκαν σε πολλά. 2003 δημόσια διζήτηση για τις ε, αποζημιώσεις ε, και λοιπά το 2006 ακριβώς και μετά αργότερα για την εξέταση αυτού του οικοσυστήματος που έχει όμως κοινοτικό ενδιαφέρον. Δεν ε, ε, μας είπαν γιατί δεν είχαν εναλλακτικές λύσεις καλύτερες για το περιβάλλον και ούτε επίσης από μια ανεξάρτητη αρχή για το περιβάλλον για όλες αυτές τις μελέτες επί των επιπτώσεων και ακόμα τα είδη που προστατεύονται και δεν εξετάστηκαν καθόλου στην δημόσια συζήτηση. Επίσης παραβίαση της οδηγίας πτηνών και του ε, ε, χώρου που οι πολίτες ζουν και επίσης η εργασία που έγινε κατά την άποψή μας δεν ήταν καλής ποιότητας και για τη βιοπικιλότητα. Η πτυχή αυτή δεν υπήρξε καμία απόδειξη ότι δεν υπήρχε καλύτερη λύση και τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι κάπως πειραματικά. Δεν είναι σίγουρα, δεν θα διαρκέσουν πολύ και είναι μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τις εργασίες που σύντομα θα ξεκινήσουν και που δεν ή δεν επαρκούν για μια κατάλληλη προστασία των ειδών που απειλούνται και για την εγρή αυτή περιοχή λέει ο αναφέρον ότι η περιοχή αυτή λέει για οροπέδιο ενώ ε, είναι με μια ειδική μορφή και καλύπτει όλο αυτό το χώρο που θα κατασκευαστεί το αεροδρόμιο. Δεν στέκει με τα υπόλοιπα που λέει η Γαλλία, ας πούμε, για το πώς ε, εξετάζεται και η οδηγία, πώς η οδηγία για τα ύδατα και πρέπει να έχουμε μια καλή ποιότητα υδάτων. Το ίδιο ισχύει όπως και για τα είδη που προστατεύονται. Όλα αυτά όμως δεν είναι κατάλληλα οργανωμένα, είναι ανεπαρκή τα έχουν οργανώσει μόνο και μόνο κατά τη διάρκεια, για τη διάρκεια των εργασιών. Σας έχουμε ορισμένες φωτογραφίες, το πώς έχει ο χώρος, βλέπετε εκεί πέρα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διάταξη, βλέπετε ένα μονοπάτι, βλέπετε τα ζώα εκεί, τα είδη κλπ. Και άλλωστε υπάρχει μια κτηνοτροφία πραγματικά που ε, είναι ιδιαίτερα παραγωγικά παραβιάζονται τουλάχιστον έξι οδηγίες κοινοτικέ. και δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες χωρίς να γίνει μια εξέταση αυτής της, αυτού του υγρότοπου. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος. Μαρή Κροντμπλίν από πλευράς Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Κριστική Επιτροπή, να σας πω ότι ναι, είχαν, είχαμε δει αυτά τα προβλήματα στα πλαίσια της αναθεώρησης της οδηγίας για τις παρεμβαντικές επιπτώσεις. Ακούσαμε τον αναφέροντα και τον ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση του οι παραστήσεις βασίζονται σε δύο στοιχεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Πρώτα απ' όλα για το περιβάλλον και επίσης για τις κρατικές επιδοτήσεις ε, βοήθειας. Και εδώ για μας ε, εδώ είναι ευκαιρία να συμπληρώσουμε τα διάφορα πληροφορικά στοιχεία για τα από την τόπου εξέταση και που τα στοιχεία αυτά και και το τελευταίο σημείο αυτής της προκαταρτικής μου παρατήρησης. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω πώς έχει το όλο θέμα ο φάκελος αυτός στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ασχοληθήκαμε με το θέμα στα πλαίσια της αναφοράς των αναφορών που κατατέθηκαν σε εσάς και ζητήσαμε από τη Γαλλία και αυτό έγινε αρχές Ιανουαρίου του 2013 στα πλαίσια τη χρησιμοποίηση αυτής της ειδική ορολογίας ε, μηχανισμός του U pilot που σημαίνει διασταυρούμενες πληροφορίες με τα κράτη-μέλη και εμείς θεωρούμε ότι Χρειάζεται να το εξετάσουμε αυτό γιατί ίσως υπάρχουν παραβιάσεις ε, του κοινοτικού δικαίου. Αυτό λοιπόν, αυτά ζητήσαμε, υποβάλαμε ερωτήσεις, κανονικά θα πρέπει να έχουμε και τις απαντήσεις. Δεν έχουν ξεπεράσει το χρονικό όριο, την προθεσμία οι γαλλικές αρχές για να μας απαντήσουν για το περιβάλλον λοιπόν. Περιμένουμε πάντα τις απαντήσεις τους. Σημειώσαμε όλα αυτά τα σημεία μετά από την ανάλυση που μας έγινε. Θα θέλαμε και πάλι να ευχαριστήσουμε τον αναφέροντα για τα κύρια σημεία που προκαλούν προβλήματα και διασταυρώνονται αυτά με τις δικές μας αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν να κάνουν και με τη μελέτη επιπτώσεων με τις οδηγίες σχεδίων και προγραμμάτων σχεδίων και επίσης τα διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την προστασία του και των διαφόρων ειδών και επίσης των πτηνών, οδηγία για τα πτηνά γιατί περιλαμβάνεται και αυτή η πτυχή αλλά είναι πρόωρο προς το παρόν να σας ε, πούμε ποια θα είναι η εκτίμησή μας ε, γιατί Εντάξει υπάρχει ένα δικαίωμα υπεράσπισης του καθένα και χρειάζεται να ακούσουμε τις, μετά από τις αναλύσεις μας τις διάφορες εξηγήσεις που θα μας δώσουν οι γαλλικές αρχές για το θέμα αυτό πάντα. Άλλωστε αυτή είναι η συνηθισμένη διαδικασία και έτσι προχωράμε στα πλαίσια και του U-Pilot. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος βέβαια Αυτήν αφορά κυρίως το θέμα, αλλά εξέφασε την επιθυμία να συνεργαστούν και συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, γιατί υπάρχουν και διάφορα στοιχεία, σημεία που έχουν να κάνουν με τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις κρατικές βοήθειες. Και στο πρόγραμμα FEDER για την περιοχή του Λουάρ Αυτά και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Μπούλαν. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ. Καταρχήν, για να είμαι συνεπής με τη σκέψη μου, να σας πω ότι λυπάμαι που γι' αυτό το θέμα αίθουσα εδώ, η οποία είναι πολύ πρόρε. Έχουμε να κάνουμε την απάντηση του γαλλικού κράτους σε σχέση με τη διαδικασία και τα συμπεράσματα της Επιτροπής για το διάλογο. Όταν μαθαίνουμε ότι δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα και σήμερα μαθαίνουμε ότι ένα θέμα είναι, ενώ είναι μερίσια διάταξη μου ζητούν να αναβληθεί θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά κοιτάξτε αν είχε, ε, υπήρξε ενημέρωση 8 μέρες νωρίτερα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή στο διάλογο εγώ είμαι υπέρ κάτι τέτοιο και θα μπορούσαμε να δούμε κάτι το οποίο γίνεται όχι και τόσο συχνά στην Επιτροπή να έχουμε μια πιο ρεαλιστική συζήτηση συγκεκριμένη για να μπορέσουν να προβληματιστούν όλοι, όλα τα μέλη της Επιτροπής να γίνει σωστή ε, διαγνωστική και να, έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής θα ήταν καλύτερα ίσως να αναβάλουμε ε, το θέμα για μια άλλη φορά. Και θα είχαμε κάτι πιο αποδοτικό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη και να δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτον, να μην συγχαίρουμε τον εθνικό, τον εθνικό διάλογο και το, με τον ευρωπαϊκό. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι βουλευτές, σεβόμαστε κάποιες οδηγίες και δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες σε ένα διάλογο που είναι καθαρά περιφερειακός ή εθνικός. Δεν είναι η θέση μας αυτή. Ο καθένας σας, Γάλλος ή όχι, Ε, προβληματίζεται και μπορεί να με ρωτήσουν για διάφορα θέματα αυτού του σχεδίου σε σχέση με τις αερομεταφορές, για την οικονομική διάσταση, αλλά εδώ στη δική μας Επιτροπή είμαστε για κάτι άλλο. Έχουμε αναφορές πάνω στις οποίες θα απαντήσουμε όταν γίνει αποδεκτή μια αναφορά. Και όταν λέω αποδεκτή, δεν εννοώ ότι την εγκρίνουμε, ότι μπαίνει στα πλαίσια τα οποία έχουν οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνει αναφορά όπου εμείς πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση και να δώσουμε μια απάντηση, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις. Έχουμε λοιπόν ένα προβληματισμό σήμερα στην Επιτροπή μας. Και, και αυτή έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Το πεδίο αυτό αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το περιβάλλον όσον αφορά το αεροδρόμιο. Και πρέπει φυσικά εδώ να δούμε τις διάφορες διαστάσεις του θέματος για το χώρο ο οποίος έχει ε, χαρακτηριστεί Natura 2000, ε, άλλες πτυχές του θέματος που έχουν φέρει η υψηλή ποιότητα για το περιβάλλον, αν έχει προβλεφθεί ή όχι από το νέο αεροδρόμιο. Επίσης το θέμα τα, της ενεργήτης κατανάλωσης ανά επιβάτη, όλα αυτά μας αφορούν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει στην Επιτροπή μας να έχουμε είναι δυνατόν πιο αντικειμενική, μια γνωμοδότηση ως δυνατόν πιο αντικειμενική και να περιμένουμε τα συμπεράσματα της Επιτροπής που είναι σημαντικά για μας και αυτά τα συμπεράσματα δεν μπορούμε να τα έχουμε αν δεν έχουμε τις μελέτες στην πιλωτική ε, ε, ε, μελέτη γαλλικό κράτος ζήτησε μια αναβολά 15 ημερών. Δεν είναι. Δεν τίποτα. Μπορούμε να περιμένουμε. Η Επιτροπή μου φαίνεται αύριο θα απαντήσει. Ε, πραγματικά. Ε, ε, θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε ένα πιο επικοδομητικό διάλογο, πολύ πιο συνεκτικό. Δεν θέλω τώρα να υπερβάλλω. Μιλάμε πολύ νωρίς και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση αυτών που κάνουν μια αναφορά. Διότι φέρπιν δεν είμαστε σε θέση να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα. Δεν με ενδιαφέρει ο εθνικός διάλογος. Θα κλείσω λέγοντας αυτό, αυτή η αναφορά να παραμείνει. Συμφωνώ αλλά να κάνουμε μια αναβολή για το διάλογο για μια άλλη ημερομηνία, όχι τόσο μακρινή, αφότου έχουμε τα συμπεράσματα και πέρσι μάλιστα ζήτησα και το ζητώ επίσημα ξανά εδώ στην Επιτροπή μια ε, έρευνα επιτόπου από την Επιτροπή Αναφορών. Επιμένω σε αυτό. Δεν θα πρέπει να μπει ε, ε, στη συζήτησή μας ο εθνικός διάλογος. Το λέω για, τους, για αυτούς που κάνουν αναφορές. Υπάρχει μια, υπάρχει μια ε, αποστολή, μια αντιπροσωπεία Φερρυπίνη, η οποία δεν περιλαμβάνει άτομα τα οποία εκπροσωπούν το κράτος το οποίο γίνεται η επίσκεψη. όλοι δεν μπορούν να πάνε το λόγο εκ μέρου αυτή τη Επιτροπής. Και, αυτή, και γι αυτό, γιατί γίνεται αυτό. Ούτω ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση ε, ευρωπαϊκή σε ένα ευρωπαϊκό θέμα και όχι να μπαίνουν μέσα οι περιφερειακές ή οι τοπικές ε, πολιτικές και αντιπαραθέσεις. Να παραμείνει δηλαδή, το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λέω λοιπόν σε αυτούς που κάνατε αναφορά να μην φοβούνται ή να μην ελπίζουν ε, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, ε αντιπροσωπεία για μια επιτόπου έρευνα θα γίνει αντικειμενικά. Επιμένω λοιπόν να συνεχίσουμε και να γίνει αφότου έχουμε τα συμπεράσματα όσο δυνατόν πιο γρήγορα ιδέουσα, ιδέουσες ενέργειες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για όσα διαφωτιστικά μας είπαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έδειξε τις ικανότητες της εδώ. Καλοθετικό είναι να τονίζουμε για την Επιτροπή ότι κάνει καλά τη δουλειά της. Δυστυχώς η γαλλική κυβέρνηση δεν είναι παρούσα με εκπρόσωπό Κρίμα γιατί θα μπορούσε να μας διαφωτίσει σε διαφορά άλλα στοιχεία, με διάφορα άλλα στοιχεία και ακόμα θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια ένταση επιτόπου και θα έπρεπε όλα αυτά να εξεταστούν ε, τάχιστα παρόλε προσπάθειες που καταβάλλονται. Παρακαλώ, συνάδελφοι, προσέξτε τα εξή τρία σημεία και να σα υποβάλω προτάσει. Ίσως υπάρξει μια κάποια, κάποιο σημείο σύγκλησης με τον συνάδελφο Μπουλάν. Διαφόρα για το σήμερα για την κατεπίγουσα εξέταση χωρίς να περιμένουμε τις διαδικασίες της U-Pilot και με την Επιτροπή Διαλόγου από το Γαλλικό κράτος, Επιτροπή Διαλόγου που, σας, που την προσκαλούμε να καταλάβει την ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του θέματος. Να το δούμε αυτό. Τι βλέπουμε ότι ε, πάντα πρέπει να είναι κάτι για να λύσει παρόμοια προβλήματα παραβίασης ε, και εμείς θέλουμε να αποφύγουμε κατάσταση που δεν θα γυρίζει πια πίσω και να αποφύγουμε επίσης και αντιδικίες που θα μας στοιχήσουν χρήμα και χρόνο. Για την Νότ Dame την περίπτωση αυτή, Εκεί διάφορα πράγματα μοιάζουν με ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε τη βδομάδα μας πέρα στο Λομέλια. Είναι το αεροδρόμιο του Βιέννα. ψήφισε κάτι το κοινοβούλιο και νομίζω ότι μετά από την περίπτωση αυτή και με άλλες περιπτώσεις που εξετάθηκαν από το κοινοβούλιο νομίζω ότι μπορούμε να λάβουμε την ευθύνη μας ε, σαν ευρωβουλευτές εδώ μέλη της Επιτροπής αναφορών και να μπορέσουμε να γνωμοτήσουμε τώρα και ακόμα για την οικονομική και νομική πτυχή. Η οικονομική πτυχή που αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και πια δούμε πού θα νομιμοποιήσει τη μην ακριβώς στήριση το δικαίωμα ότι αυτά τα όσα έχουν να κάνουν με τις οικολογικές επιπτώσεις όλα αυτά τα πράγματα αλλά προσέξτε όλα αυτά δεν είναι καθόλου αντικειμενικά είναι μια εκτίμηση πανάρχια, σκουριά Κοιτάξτε και το κόστος αυτού του σχεδίου απέναντι σε υποθετικό όφελος. Κοιτάξτε το κοινωνικό κόστος, το εργατικό κόστος, εκεί κάτι εκεί, το περιβάλλον, το κόστος του περιβάλλον. Μια και ο υγρότοπος αυτός δεν θα διαφυλαχτεί. Οικονομικό, Δηλαδή 500 εκατομμύρια δημόσιο χρήμα που θα μπει εκεί. Είναι το δημόσιο χρήμα των πολιτών. Και είναι ένας υγρότοπος που με το ρόλο το σημαντικό που παίζει και για να υπάρχει πάντα νερό και ακόμα για τα διάφορα σημεία όλα αυτά που θα αποβούν εις μας και δεν υπάρχει επιστροφή. Και εδώ το 2013 βλέπουμε ότι περισσότερα θα μας κοστίσει παρά να μας ωφελήσει. Και το 1960 μιλούσαμε για μεταφορά δρομίων. Τώρα μιλάμε για ένα νέο αεροδρόμιο κάπου σε μια περίπου υπάρχουν 14 δρόμια. Νέο αεροδρόμιο που δεν μπορεί να συμφιλειωθεί να συνδυαστεί με τους δικούς μας στόχους. Προπολά κατά του κλίμακος, της διευκαιοπικιλότητας, όλα αυτά τα πράγματα και θα μην ξεχνάμε και την αύξηση του κόστου των υδρογονανθράκων. Και κάτι ακόμα και ολοκληρώνω Παρόλο που οι δύο αναφορές, δύο εκεί είχαμε, είχαν τους καλύτερους νομικούς από πλευράς Γαλλίας, τους ειδικού και με πολλές καταδίκες της Γαλλίας επειδή δεν σέβεται αυτό το δίκαιο το κοινοτικό. Συνάδελφοι, εάν εντάξει για να αποσχηματίσετε πλήρη ε, άποψη για αυτή την παραβίαση, για το περιβάλλον, αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέραμε, την οδηγία για τα σχέδια, τα προγράμματα, είτε για την ύδατα, είτε για το περιβάλλον. Αν θέλετε να περιμένετε τη νομική ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των απαντήσεων της γαλλικής απάντηση από το γαλλικό δημόσιο, τότε θα ήθελα να σα προσκαλέσω κάτι. Ρίξτε μια ματιά ότι υπάρχει πραγματικά αμφιβολία επί τόπου η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί για να ε, μην μπορεί κανείς να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση ε, επιταχύνει τις και επίσης χρησιμοποιεί και στρατό για την προστασία χωρίς να υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε υπεύθυνοι σαν ε, ευρωβουλευτές και αυτό στους Γάλλους πολίτες και στην κυβέρνηση να απευθύνουμε αυτό το μήνυμα. Εμείς είμαστε επί τόπου, έχουμε σχέση με το χώρο, με τον τόπο και δεν δεχόμαστε ένα παρόμοιο σχέδιο που είναι αντίθετο με τις αξίες, με το περιεχόμενο αυτών που εμείς ψήφισαμε στο Κοινοβούλιο, δημοκρατικά και περιβαλλοντικά. Προτείνω και να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, αλλά για να δούμε και το πώς έχουν τα πράγματα. Παρακαλώ, όπως ο κ. Μπουλάν είπε, να αποστείλει μια αντιπροσωπεία με επίσκεψη εκεί των αεροδρομίων που υπάρχουν ήδη, να συναντηθούν με το, το προσωπικό, να δούμε τι γίνεται, ποιες αντιδράσεις υπάρχουν, να δούμε τους φυσικούς ε, πόρους πήγες τόπους και επίσης εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στείλουμε μια επιστολή στο γαλλικό κράτος, στη γαλλική κυβέρνηση να διακόψει οποιαδήποτε εργασία εκεί από τη στιγμή που αυτή η εξέταση δεν θα έχει τερματιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, ίσως αυτό το σχέδιο θα μπορούσε έτσι να διακοπεί χωρίς δικαστικές προσφυγές και έτσι θα έχουμε βοηθήσει και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουν παρουσιαστεί σχεδόν όλα τα επιχειρήματα να επενθυμίσω. Να πω ότι δεν έχει γίνει ακόμα η θεμελίωση ε, του αεροδρομίου. Έχει ξεκινήσει μεν. Είναι σημαντικό όμως να δούμε όταν να δούμε όταν ορισμένες ε, το, αρχές μπαίνουν σε μια ε, σιγουριά όταν ξεκίνησε αυτό το σχέδιο ε, από, από την αρχή ε, όλες οι εναλλακτικές λύσεις είχαν απορριφθεί. Από τη στιγμή πολιτικά εγκρίθηκε αυτό το σχέδιο, πριν ακόμα να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος, υπήρχε υπήρξε μια τάση να αναγνωριστεί ότι τόση σημαντική χρησιμότητα αυτού του σχεδίου που θεωρήθηκε ότι μπορούν να καταστραγηθούν όλες οι άλλες οι ευρωπαϊκές αρχές. Παραπληροφόρηση, ε, προσπάθεια να φανεί ότι ε, αποφασίστηκε, θα ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, αλλά ένα κράτος πρέπει να σεβασεί ε, κάποιες αρχές, κάποιους κανόνες. Υπάρχει το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον και είναι αυτό το οποίο διακυβεύεται. Ευχαριστώ. Thank you, η κυρία Ζανόκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μου η παρέμβαση είναι ανάμεσα από αυτές των εκπροσώπων από τη Γαλλία. Είδαμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες της διαφάνειας. Εγώ είμαι από την κεντρική Ευρώπη, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στην Γαλλία υπάρχουν τόσο πολύ όμορφα μέρη. Από την κεντρική Ευρώπη, συγγνώμη, και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στην Γαλλία υπάρχουν τόσο όμορφα μέρη. Είναι μία από τις αρχές μας η διατήρηση της φύσης και το ΕΛΚ χρησιμοποιεί ορολογία πρασίνων πια για την, το πρασίνισμα της ανάπτυξης κτλ. Δεν νομίζω όμως ότι αυτές οι λύσεις ακολουθούν αυτή την άγουσα. Γι' αυτό εξετάζουμε αυτή την κατάσταση τώρα. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορεί να διορθωθεί είναι μία αναστρέψιμο. Ε, προσπαθούμε να αναστρέψουμε κάτι μία αναστρέψιμο. Υποστηρίζω την πρόταση να γίνει διερευνητική αποστολή. Πήγαμε και στη Γαλλικία πρόσφατα και είδαμε ότι κάποιες αποφάσεις είναι μη αναστρέψιμες και δεν ξέραμε πώς να τις διαχειριστούμε. Οπότε αν έχουμε μία ε, δυνατότητα να σταματήσουμε αυτή την θεωρούμενη ως λύση που μπορεί να καταστρέψει αυτή την προστατευόμενη περιοχή που ανήκει και στις προστατευόμενες περιοχές των οδηγιών της Ένωσης, τότε ας το πράξουμε. Υπήρξε, έγινε και η κατασκευή ε, ενός, ε, ε, μιας πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου που κατέστρεψε ε, κάποιους ε, βιοτόπους πουλιών και δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις πολλών δεν σταμάτησε η κατασκευή. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε στη Γαλλία α, τους ανθρώπους αυτούς που έχουν υποβάλει την αναφορά. Εγώ προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, να κάνουμε μια διαρευνητική αποστολή και να περιμένουμε να δούμε πιο εις αξιολόγηση και να ακούσουμε βέβαια και τις απαντήσεις της γαλλικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αγαπητοί αναφέροντες, αγαπητοί φίλοι, εδώ πρόκειται για ένα γαλλογαλλικό εμφύλιο πόλεμο. Ναι, λυπάμαι, λυπάμαι πάρα πολύ που ένα τόσο σημαντικό και λεπτό ευαίσθητο θέμα εκεί βλέπουμε και ένα τίμημα πολιτικό κάπου χωμένο ανάμεσα. Και άλλοι συνάδελφοι συμμερίζονται την άποψη αυτή. Τώρα, για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση που είναι απαραίτητε αυτές τώρα αυτή την εποχή κρίση ακόμα περισσότερο και το πώ επηρεάζεται η κατάσταση όχι μόνο στην Ονταμπτελάντ, αλλά και σε όλη την περιοχή και τι θα πρέπει να γίνει σεβαστό από πλευρά περιβάλλοντο. Όλα αυτά που μας απασχολούν θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς πάνω σε αυτά. Οι αναφορές να παραμείνουν ανοιχτές για να έχουμε μια σαφή συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα, να έχουμε από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές επίσης μια απάντηση και με τις δύο αυτές θέσεις απαντήσεις και από τη στιγμή που και εκείνοι και οι αναφέροντες ε, ενδιαφέρονται πάντα να μπορέσει να ζητεί το θέμα σε επόμενη συνάντηση και μάλιστα εάν κριθεί απαραίτητο να πάμε επί τόπου να δούμε πως έχει κατάσταση για να μπορέσουμε να λάβουμε απόφαση να πάμε στην Ονταμντελάντ για να δούμε επί τόπου τα γεγονότα. Μη συγχωρείτε και για τα γαλλικά μου, τέλος πάντων προσπάθησα. Και Βλέπουμε ένα πολιτικό πάθος, σχεδόν φανατισμό και θα πρέπει να είμαστε αντίθετα ρεαλιστές, να βασιστούμε στους νόμους. Εγώ σέβομαι ιδιαίτερα τους γαλλικούς νόμους και να σεβαστούμε και την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη δυνατότητα έκφρασης κρίσης. Ευχαριστούμε. Κανέκ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και εγώ τους αναφέροντες για την ποιοτική παρουσίασή τους, στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή και την Επιτροπή Αναφορών. Δεν ανήκω εγώ, αλλά όπως συνάδελφος Αντριμπελιέ, εγώ λυπάμαι γιατί είναι απούσα η γαλλική κυβέρνηση με ένα εκπροσωπό της. Εσείς εκεί ανήκετε και υποστηρίζετε η πολιτική σας ομάδα. Όχι, όχι, όχι εσείς προσωπικά, εντάξει. Αλλά λυπάμαι για την απουσία αυτή. Είμαι και Γάλλος βουλευτής και από τη Βρετάνη ταυτόχρονα λοιπόν στο αεροδρόμιο Νόρα Ατλαντικ. το χρησιμοποιώ συχνά αυτό το αεροδρόμιο και διαπιστώνω συχνά ότι ε, υπάρχει τρομερή κίνηση εκεί. Ήδη είχαμε μακρές συζητήσεις, πραγματοποιούνται πάντα συζητήσεις, τα δημοκρατική διαδικασία. Αλλά οι περισσότεροι εκλεγμένοι της ε, Βρετάνης και του Πεντελουάρ εκφράστηκαν υπέρ του σχεδίου αυτού, τουλάχιστον η πλατιά πλειοψηφία. Και εκ μέρους τους ε, λέμε ότι απαιτείται η είδηση αυτού του αεροδρομίου. Και ο κ. Μουστιέ το είπε μια παρατήρηση χωρί χωρίς ε, μικρόφωνο δεν ακούμε δυστυχώ. Μισό λεπτό λέω ο μιλητής να ολοκληρώσω. Όχι, δεν θα στην οικονομική πτυχή. Ας πω τι με απασχολεί περισσότερο. Το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν είναι αποκλειστικότητα ορισμένων μόνο ε, Αφορά τη δεξιά, την αριστερά, το κέντρο, εντάξει και ε, είμαστε επί τόπου μας αφορά. Και να σας πω και για την ε, βιοπικιλότητα ας πούμε και για την ε, προστασία του υγρότοπου, τη διατήρησή του. Ξέρετε ότι εγώ επιμένω ότι γνωρίζω πολύ, ιδιαίτερα αυτά τα θέματα γιατί είμαι επιτόπου και ειδικό και διευθύνων ε, της ε, υπηρεσίας Σιδάτων. Και εκεί, επί τόπου έχουμε υπεύθυνο κόσμο που εργάζονται, που είναι από τους πολίτες, από τις μη κυβερνήσεις από τους γεωργούς και όλοι αυτοί είπαν ναι για το σχέδιο. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι συμμετέχει εκεί σε αυτή τη πλησιδά τον κόσμο υπεύθυνο. Και θα πρέπει να δούμε για την ενδεχόμενη καταστροφή του υγρότοπου, να δούμε τι προβλέπεται από την οδηγία για τα ύδατα. Δεν νομίζω λοιπόν, πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίθεση. Αυτό που είπε ο ήταν πολύ καλά και ωραία. Είναι ιδεολογική γαλλογαλλική συζήτηση, κρίμα. Συμφωνώ με αυτό. Ελπίζω ότι η λογική θα κερδίσει τη μάχη και να σας πω ότι είμαι υπέρ της άποψης του αδερφού Μπουλάν και της πρότασής του. Να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες τις τωρινές και μετά γιατί όχι, ξώμας επιτροπής, να οργανώσουμε ένα ταξίδι επιτόπου στη Βρετάνη, να βάλουμε και σε αδιάφορες μπότες μας για να πάμε να δούμε τα πράγματα εκεί στον υγρότοπο. Αυτά για να δούμε τι ευσταθεί και τι όχι από όλα αυτά που υποστηρίζονται εδώ. Ευχαριστούμε ο Μποβέ, κύριος Μποβέ. Σας ευχαριστώ που από την Επιτροπή Γεωργίας υποδέχεστε εμένα Ευρωβουλευτή, δεν θα επισέλθω στην τοπική εξέταση του θέματος. Καταλαβαίνω τόσο ο κ. Κατέκ ότι θέλει να πάει κοντά κοντά εκεί που μένει ο ίδιος 50-60 χιλιόμετρα. Εντάξει, αστείακι, αστείακι, αστείακι είπα ε, ότι θέλετε να έχετε αεροδρόμιο στα πόδια σας, δίπλα σας. Έχει χάσει το δικαίωμα να κάνει και αστείακια και επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία και επειδή διαθέτω και μια κάποια πείρα. Ε, ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Αλλά με την πείρα μου έχω καταλάβει ότι σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Το γαλλικό κράτος ε, έχει ένα πρόβλημα με τη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι αποφάσεις κοινή ωφέλεια. Είναι πρόβλημα αυτές οι αποφάσεις και είναι μια προστασία κρατική πολύ συχνά ενάντια στους πολίτες και όχι από την άλλη μεριά από τους πολίτες απέναντι στο κράτος και θα πρέπει να δούμε μέσω μιας δημοσυζήτησης πώς θα ευθυγραμμιστεί το κοινοτικό δίκαιο με το εθνικό δίκαιο. Σας το λέω επειδή ήμουν επιτόπου εκεί όταν το 1971, λοιπόν πάνω από 40 χρόνια πριν, ε, 103 οικογένειες στις 14.000 εκτάρια ε, αποφασίστηκε να εκδιωχθούν αυτοί οι κάτοικοι εκεί για μια εγκατάσταση στρατιωτική και κέρδισαν τελικά αυτές οι 103 οικογένειες. Και τώρα 40 χρόνια μετά οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης λένε ότι ναι ήταν λάθος αυτός ο σχεδιασμός να τους διώξουν τότε και ευτυχώς που κέρδισαν οι κάτοικοι. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα όσον αφορά τον τρόπο λήψη αποφάσεων. Λοιπόν, η ερμόνιση του εθνικού με το κοινοτικό δίκαιο έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αλλά τι γίνεται, η όλη διαδικασία η δικιά σας ε, της Επιτροπής Αναφορών με την Επιτροπή, με το γαλλικό κράτος. Έτσι όμως ενδεχόμενα θα μπορούσαμε να δούμε και μια διέξοδο από μια μεριά ή από την άλλη. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ξέρετε κανονικά ποια είναι η θέση μου έτσι, αλλά επαναλαμβάνω δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προχωράμε ένα σχέδιο από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η όλη εξέταση του θέματος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ότι το δικαίωτο κοινοτικό το ευρωπαϊκό θα πρέπει να υπερισχύσει του τοπικού, οικονομικού κλπ. κλπ. Άρα λοιπόν έχουν δικαίωμα να επικαλεστούν αυτό οι Γάλλοι κάτοικοι που αντιδρώνουν. Ναι. Ε, ε, λοιπόν, παίρνω το λόγο. Κοιτάξτε. Ε, συγχαίρω και εγώ αυτούς που κάνατε αναφορά και ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Αλλά να πω δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο διάλογος θεωρείται γαλλογαλλικός. Ε, μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο ε, είναι, θα γίνει διεθνές. Στην Ευρώπη χρειάζεται εδώ και εκεί να κάνουμε οικονομικές επιλογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε γαλλικό. η επιλογή είναι ανάμεσα στο σιδηρόδρομο και το αεροδρόμιο πρέπει να γίνουν ανάλογε ε, ε, οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε και να καταλάβουμε ποια είναι αυτό που, είναι, που μας συμφέρει. Προσοχή όμως, αυτό που διακυβεύεται είναι, δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται στη Γαλλία. Ξεπερνάει τα γαλλικά σύνορα. Πέρα από τους γεωργούς επιτόπου υπάρχουν πολλοί νέοι που φτάνουν σε αυτή την περιοχή για να ζήσουν και είναι από άλλες ε, εθνικότητες. Τώρα, αν αφήσουμε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση να επιβάλλει κάτι και σε άλλες περιοχές το είδαμε στη Γαλλία με αρνητικές επιτόσεις να σας αναφέρω τι έγινε Φερρυπίν στο Σούπερ Φίνικα στη δεκαετία του 70. Οι επιπτώσεις ήταν αρνητικές, υπήρχαν νεχροί και από τις δύο πλευρές. Θεωρώ η Επιτροπή για τις αναφορές πρέπει να στείλει μια αντιπροσωπεία ώστε να τον πιο γρήγορα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της φυσικά. Είναι απαραίτητο κατά με διότι τα στοιχεία που έχω εγώ από όλου, όσοι, όσους αφορά, γεωργούς ε, και λοιπά και φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας ε, θέλει να επιβάλλει βιαίως θα λέγαμε κάτι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ένα λεπτό. Λιγότερο λέει ο μιλήτρια. Δεν είναι γαλλογαλλικός διάλογος. Εμείς είμαστε ευρωβουλευτές εδώ. Υπάρχουν κείμενα της Ευρώπης που καταστρατηγούνται σήμερα εν δυνάμει. Ε, έχουμε με κείμενα που αφορούν τα, τα ύδατα και Τα, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Εμείς θα πρέπει να δούμε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συμφέροντος και οι αποφάσεις που λαμβάνουν σε εθνικό επίπεδο. Ε, δεν είναι το πρόβλημα πώς, για τους μεν και τους δε που θέλουν να αποφασίσουν κάτι. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο για το επίγον του θέματος. Σήμερα να αποφασίσουμε για μια επιτροπή ερεύνης επιτόπου όλα μας δείχνουν ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία και ότι το γαλλικό κράτος θέλει να επιβάλλει βίαιος κάτι. Θα πρέπει να πάμε εκεί να δούμε. Να δράσουμε δηλαδή όσο είναι καιρός. Να δείξουμε στους Ευρωπαίους και Γάλλους πολίτες ότι μπορούμε να δράσουμε γρήγορα και να εμποδίσουμε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Ένα λεπτό ο καθένας για την απάντηση, έτσι, και για τους ε, αναφέροντες. Παρακαλώ, κυρία μου, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε εδώ σήμερα. Ίσως ήταν πρόωρο για ορισμένες. Δεν περιμένα βέβαια μία απάντηση για το αν χρειάζεται ή όχι αυτό το αεροδρόμιο εκεί. Αλλά θέλαμε να σας κάνουμε να προσέξετε ότι είναι κατεπήγον να μην προχωρήσουν οι εργασίες, να μην ξεκινήσουν πράγματα και να γίνει μη αντιστρέψιμη, να μην μια αντιστρέψιμη κατάσταση. Μη αντιστρέψιμη. Ναι, περιμένουμε την γαλλική απάντηση και σε όλα αυτά τα ερωτηματικά που αναφέρατε. Ναι, δεν διεξάγεται μια γαλλογαλλική πολιτική συζήτηση γιατί ο καθένας βλέπει τα πράγματα από διαφορετικές ε, πτυχές. Και εδώ, εδώ είναι ο δήμαρχος του περιοχής και εγώ είμαι υπεύθυνη εκεί και ξέρω ότι το αεροδρόμιο που λένε ότι δήθεν είναι κορεσμένο ε, δεν είναι κορεσμένο, το ξέρω απέθυνα. Ναι, εγώ θα ήθελα να σας το εξή. Η συμμετοχή νομικών από όλη τη Γαλλία που είναι δικευμένη στο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο γιατί ενδιαφέρονται. Θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα και το ε, κάνουν ε, βασιζόμενοι σε ένα κείμενο που θα πρέπει να σε γίνει σεβαστό ιδιαίτερα για να υπάρξει μια διαφορετική οικονομική σε αυτές τις περιοχές και προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω κάτι θέμα χωροταξίας, οργάνωσης, ε, μακριά από τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα και αυτό το αεροδρόμιο βοηθάει στην ανάπτυξη οικονομίας. Με βιομηχανική δραστηριότητα και τα ενδιαφέρουσα. Επίσης η Airbus με 20.000 άμεση έμεσες θέσεις εργασίες οργάνωση πολύ σημαντική και οικονομικά, κοινωνικά και βέβαια και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα πράγματα μπαίνουν στο παιχνίδι της εξέτασης ε, για να δούμε τις προτεραιότητάς μας. Και το λέω, επιμένω, τι θα είναι μερικοί να βάλουν ε, κάτω από ένα γυάλινο κόδωνα την περιοχή εκεί. Χρειαζόμαστε μια κινητικότητα, χρειαζόμαστε να έχουμε επαφή με τις μεγάλες αγορές ε, και με το αεροδρόμιο του Notre Dame de Εκεί θα είναι το μελλοντικό μας αεροδρόμιο και ακριβώς αυτό το στόχο θα εξυπηρετήσει. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να παρατηρήσουμε, αλλά είναι επίγον να, ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Εφιστούμε την προσοχή επίσης ότι ε, θα πρέπει να δείτε το θέμα του σεβασμού της οδηγίας διότι το γαλλικό κράτος δεν έχει πράξει σωστά και θα υπάρξουν επιπτώσεις στη, στη, στη, στη στο, στην περιοχή μας σε σχέση με τη δημιουργία αυτού του αεροδρομίου όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω παρεμβάσεις. Είμαι με τον κύριο Μιστιέρ. Είμαι πρόεδρος στην περιοχή, τη μετροπολιτική περιοχή της Λαντ και είμαι από μια ε, κοινότητα πάνω από την οποία περνάνε τα αεροπλάνα και υπάρχει το πρόβλημα του θορύβου. Εγώ μπορώ να σας πω ότι τοπικά στην περιοχή της Νάντης και ο... Ε, η μεταφορά του αεροδρομίου θεωρείται αναπόφευκτη. Κάθε μέρα τα αεροπλάνα περνάνε πάνω από το κεφάλι μας. Υπάρχει ανησυχία από, του από τους κατοίκους και υπάρχουν περιορισμοί οι οποίες μας εμποδίζουν να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό που έχουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσετε ήρεμα όλα τα δεδομένα και να, δείτε ότι ε, να γίνει χρήση ώστε να τον λιγότερου εδάφους και όσο να τον λιγότερου ε, υγροτόπου. Δεν θα πρέπει να, καταστρα... Δεν πρέπει να καταστραφούν και άλλες ε, περιοχές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε όλους και τους ε, υπογράφοντες την, σαν την αναφορά γιατί παρουσίασαν το θέμα αυτό και όπως είπε ο κ. Μπουρλάν μπήκε στην ημερήσια διάταξη σύμφωνα με την τακτική διαδικασία λοιπόν ε, όχι λόγω κατεπήγοντος ε, λυπάμαι που δεν το προσέξατε αυτό είχε προταθεί στην προηγούμενη συνάντηση στους συντονιστές, άρα λοιπόν εγκρίθηκε την προηγούμενη φορά, το μήνα μας πέρασε από τους συντονιστές και μπήκε στην ημερήσια διάταξη. Και σήμερα τι θελήσαμε, θελήσαμε να ακούσουμε όλους εκείνους που υπέγραφαν την αφορά αυτή και βλέπαμε, είδαμε μια πλατιά συζήτηση γιατί ακούσαμε και θέσεις υπέρ και θέσεις κατά και νομίζω ότι διανύσαμε ένα κάποιο κομμάτι του δρόμου. Ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας είπε ότι όλα αυτά που έφυξαν οι αναφερόμενοι με τις περιγραφές τους είναι σημαντικά στοιχεία για να σχηματίσουμε μια πλήρη γνώμη τουλάχιστον πληρέστερη και περιμένουμε και τις απαντήσεις της γαλλικής, των γαλλικών αρχών που ελπίζουμε να έρθουν εμπρόθεσμα. Τώρα όλοι όλοι ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή, οι αναφορές αυτές γιατί Θα πρέπει να εξεταστούν αυτά καινούργια σημεία για να δούμε λοιπόν θα ελέγξουμε τι γίνεται με τις προθεσμίες για να υπάρξουν και απαντήσεις από τις γαλλικές αρχές στην Επιτροπή και θα μπορούσαμε να παρέμβουμε και άμεσα ζητώντας οι ίδιοι από τις αρχές από όποιες δεν απαντούν εμπρόθεσμα να μας απαντήσουν. Και να το πω αυτό και προσωπικά ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που η δική μας Επιτροπή Αναφορών μπορεί να το συζητήσει πριν να έχουμε τετελεσμένα γεγονότα για ενδεχόμενα παραβίαση σημαντικών οδηγιών κοινοτικών, άρα λοιπόν παρόμοιες ε, συζητήσεις ε, αντιστοιχούν σε προσδοκίες ε, των Ευρωπαίων πολιτών που Γι' αυτό ακριβώς απευθύνονται σε μας. Παραμένουν ανοιχτέ οι αναφορές και ελπίζουμε τις γαλλικές απαντήσεις και μετά θα μπορέσουμε ίσως να οργανώσουμε και μια αποστολή μιας αντιπροσωπείας που εξετάσει επιτόπου την κατάσταση αυτά και ευχαριστώ τους υπογράφοντες τις ε, αναφορές αυτές. Το σημείο 15 τώρα είναι η αναφορά της Μισελ Τιού, Βρετανικής Ιθαγένειας, για την κατάργηση των πειραμάτων για καλλιντικά σε ζώα. Η αναφέρουσα. Παρακαλώ οι υπόλοιποι της προηγούμενης, ε, των προηγούμενων αφορών να εξέλθουν σιωπηλά για να μπορέσουμε να εργαστούμε στην επόμενη αναφορά.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 Ευχαριστώ την Επιτροπή που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε την αναφορά μας. Κέιτι Τέιλορ ονομάζομαι, εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για, την, για το τέλος των ε, πειραμάτων. Ε, εκπροσωπούμε διάφορες οργανώσεις σαν την Ευρώπη. Είμαστε ένα από του εμπλεκόμενου φορεί με του οποίου συνδιαλέγεται το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Η αναφορά την οποία σα έχουμε αναφέρει περιλαμβάνει περίπου μισό εκατομμύριο υπογραφέ και ζητά από το Κοινοβούλιο να να εφαρμόσει την 7η ε, οδηγία για τα καλλιντικά και την απαγόρευση που υπάρχει εκεί. Οι υπογραφέ λένε ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν πλέον καλλιντικά διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, γίνονται πάνω στο οποίο γίνονται δοκιμέ σε ζώα. Ικανοποιηθήκαμε πάρα πολύ από την, από την αναφορά του Επιτρόπου Μπόργκ το, ότι αυτή η απαγόρευση διάθεση στην αγορά θα εφαρμοστεί την συγκεκριμένη οδηγία που, τη συγκεκριμένη ημερομηνία που έπρεπε και δεν θα υπάρξει αναβολή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για όλο τον κόσμο. Ότι δεν είναι πλέον αποδεκτό να υποφέρουν τα ζώα ώστε να δημιουργούνται και να παρασκευάζονται καινούργια καλλιντικά. Ε, μιλούμε δηλαδή και για ε, μια απαγόρευση που ε, έχει φτάσει μέχρι και την Αμερική, μέχρι την Κίνα. Η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της απαγόρευσης ως προς αυτό. Και η αναφορά μας εξακολουθεί να υφίσταται γιατί υπάρχουν κάποια σημαντικά σημεία, κάποιες λεπτομέρειες για το πεδίο εφαρμογή απαγόρευσης που θα πρέπει να οριστεί πιο συγκεκριμένα. Και θα ήθελα να κάνω μια περίληψη των θεμάτων που μας απασχολούν ως προς αυτό. Ε, κάθε μία από τις απαγορεύσεις στον κανονισμό για τα καλλιντικά ε, αναφέρεται με, τις, ε, με τους όρους δοκιμές και τους σκοπούς αυτής της οδηγίας. Τι σημαίνει αυτό. Στην ανακοίνωσή του προς το, προς, προς το, Συμβούλιο και προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν λέει ότι η απαγόρευση αφορά ένα συστατικό όταν αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατασκευή καλλιντικών συστατικά λοιπόν που χρησιμοποιούνται κυρίως στα καλλιντικά πρέπει να ε, δοκιμάζονται με, σύμφωνα με άλλη νομοθεσία, ε, όπως ας πούμε το REACH, ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή καλλιτικών. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν αυτές οι απαγορεύσεις από μια πολύ στενή, πολύ αυστηρή ερμηνεία του όρου testing, του όρου δοκιμή για, τις, για τους σκοπούς της οδηγίας. Αυτή λοιπόν η αυστηρή ερμηνεία δεν είναι αυτή που ήθελε το Κοινοβούλιο, όπως αναφέρει και ο Γενικός Αγγελέας σε μια υπόθεση του 2000 2004. Η θέση του ήταν ότι οποιοδήποτε, ε, οποιοδήποτε συστατικό δοκιμάζεται σε άτομα, ε, σε ζώα, συγγνώμη, σε οποιαδήποτε νομοθεσία δεν μπορεί να ε, χρησιμοποιείται για τα καλλιντικά. Βέβαια, κάθε συστατικό δοκιμάζεται για διαφορετικού σκοπού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα καλλιτικά, αλλά το κοινό δεν θα πρέπει να παραπλανάται. Και δεν θα πρέπει να νομίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τις δοκιμές σε ζώα για τα καλλιτικά. Οπότε, αντί να μιλούμε μόνο για αποκλειστική χρήση, να λέμε για χρήση κυρίως στα καλλιτικά. Αυτό συνδυάζει και την θεωρία αλλά και την πράξη. Και επίσης ανησυχούμε για το ότι η Κομισιόν λέει ότι τα δεδομένα για, τα, για, τις δοκιμές αυτές σε σχέση και με τους κανόνες που επισχύουν σε τρίτες χώρες, αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα, στα ενημερωτικά σημειώματα των καλλιτικών. Νομίζουμε όμως ότι αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και στις εταιρείε. Ότι αν ένα συστατικό ε, ε, περνάει υποδοκιμή για μια τρίτη χώρα, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον στην Ευρώπη. Γιατί αυτό ακριβώς λέει και ο κανονισμός για τα καλλιτικά. Κλείνοντας λοιπόν, καλωσορίζουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν να διατηρηθεί ε, η απαγόρευση για τις δοκιμές και τη θέση σε εμπορία, αλλά ε, πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά έτσι ώστε να τηρηθεί η πρόθεση του ε, Κοινοβουλίου όταν ψήφισε τις απαγορεύσει αυτές το 2003. Προτείνουμε λοιπόν η Επιτροπή Αναφορών να παραπέμψει αυτή την αναφορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για συζήτηση, για να μελετήσει αυτές τις ε, λεπτομέρειες και να, είναι, να εξασφαλίσουμε ότι η πρόθεση του Κοινοβουλίου όταν νομοθετεί για αυτές τις ε, ε, όταν νομοθετεί για αυτές τις απαγορεύσεις θα γίνεται σεβαστή η απόφασή του. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας παρουσιάσετε την αναφορά σας. Η Κομισιόν θέλει το λόγο thank you very much. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Νομίζω ότι η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν ε, έχει έρθει στην ε, Επιτροπή σας για, το τέλος των, για την πάυση των δοκιμών σε ζώα, όπου διατηρείται η απαγόρευση για τις δοκιμές σε ζώα. Η ECIE είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός εταίρος σε όλη αυτή τη διαδικασία και έχει συνεργαστεί με την Κομισιόν πολύ στενά. Βεβαίω έχουμε συνεργαστεί και με άλλου από την Κομισιόν με τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα την ουσία, η οδηγία για τα καλλιτικά προβλέπει το phasing out των δοκιμών για τα, σε ζώα για τα καλλιτικά και οι διατάξει για τι οποίε μιλούμε τώρα εισήχθησαν το 2003 στο νομικό πλαίσιο. Τα, οι δοκιμέ σε ζώα ήδη απαγορεύονται από το 2004 για, για τα συστατικά ήδη από το 2009 και για, από τον Μάρτιο του 2009 απαγορεύεται να τίθενται σε εμπορία καλλιντικά και τα συστατικά τους εφόσον έχουν ε, δοκιμαστεί σε ζώα για να πληρούνται οι σκοποί της οδηγία Και για την θέση σε εμπορία επίσης ε, ισχύει η απαγόρευση και για τα καλλιτικά και για τα συστατικά. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχε διευρύνει την ε, ημερομηνία αυτή για το 2013. Η Κομισιόν επίσης ε, χρειάστηκε να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για, τους, ε, για το ότι ε, αυτά, κάποιες από αυτές τις δοκιμές δεν θα γίνονταν ε, μέχρι το 2013 που ήταν η προθεσμία και όπως λέει το κείμενο ζητήθηκε να υπάρξει μια νομοθετική πρόταση. Για να τηρήσουμε λοιπόν αυτέ τι διατάξει, η Κομισιόν ήδη έχει υποβάλει την αναφορά τη στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2011 ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ και συνέχισε τη δουλειά της με μια αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών σε σχέση με τούτη την προθεσμία ώστε να δούμε αν μπορούμε να την τηρήσουμε ή να την αναβάλουμε. Και επίσης σκεφτήκαμε και μια εξαίρεση. Αυτό αναφέρεται και, σε αυτό αναφέρθηκε και η αναφορά. Από την ώρα που υπευλήθη αυτή η αναφορά τον Νοέμβριο του 2012, η Κομισιόν έχει λάβει συγκεκριμένη θέση επί τη προθεσμία και έχει επιβεβαιώσει ότι προτίθεται να την διατηρήσει ω έχει, να μην κάνει πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λοιπόν. Και όπως αναφέρεται, η Κομισιόν έχει ε, υιοθετήσει στις 11 Μαρτίου, μάλλον, έχει, θα υιοθετήσει στις, ε, έχει συγγνώμη, 11 Μαρτίου μια ανακοίνωση ε, για το, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που, δια, που λέει ότι διατηρεί την πρόθεσή της να τηρήσει την προθεσμία, να εφαρμόσει την απαγορεύση και να ε, στηρίξει την έρευνα και την κοινοτομία στον τομέα αυτό. Και βεβαίως μιλούμε και για την συνεργασία με τρίτες χώρες. Θεωρούμε λοιπόν ότι με τούτη την ανακοίνωση έχουμε λάβει μια σαφή θέση και δίνουμε τις, ε, την απαραίτητα χέγγια ότι θα διατηρηθεί η απαγόρευση. Επίσης τονίζουμε την ε, κατανόηση της Κομισιόν για το τι σημαίνει η απαγόρευση. Ε, βεβαίως το δικαστήριο είναι αυτό που θα δώσει τις περαιτέρω πληροφορίες, τις περαιτέρω λεπτομέρειες. Ευχαρίστω να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και να συμπεριλάβουμε βεβαίω και άλλου εμπλεκόμενου φορεί στι συζητήσει μα, έτσι ώστε να υπάρξει συνεκτική εφαρμογή αυτή τη απαγόρευσης και βεβαίως όπου μπορούμε να συνεργαστούμε θα συνεργαστούμε με όλους όσους εμπλέκονται. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα σύντομα να πάρω το λόγο για αυτή την αναφορά, την οποία υποστηρίζω. Αυτά που λέει η Κομισιόν είναι ε, πραγματικά επί τον τύπο των ήλων για την ανακοίνωση του 2013 και για τη σχετική ε, προθεσμία για την απαγόρευση. Είναι καλά λοιπόν τα νέα. Είναι σαφής η βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, τα... Οι δοκιμές των καλλιτικών που γίνονται στα ζώα να μην γίνονται πια αποδεκτές και αυτό φαίνεται και από τον τεράστιο αριθμό υπογραφών που συνοδεύει αυτή την αναφορά. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποφέρει απλώς και μόνο για να έχουμε μια νέα ενυδατική κρέμα ή ένα νέο κραγιόν. Στον υπόλοιπο κόσμο βέβαια, οι 8 στις 10 χώρες δεν έχουν ε, τέτοιες δοκιμές που δεν γίνονται σε ζώα. Επομένως θα ήθελα αυτή η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και να προσπαθήσουμε να βρούμε περαιτέρω πληροφορίες από την Κομισιόν κυρίως για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτές τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ένα αντίστοιχο καθεστώς απαγόρευσης για, την, ε, για δοκιμές ζώα και να δούμε πώς μπορούμε να τις ενθαρρύνουμε να το διαμορφώσουν και ταυτόχρονα να δούμε και τα σχόλια το, της αναφέρουσας για να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τόσο απαιτεί η οδηγία. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το θέμα αυτό και θα μπορούσαμε να το διευκρινίσουμε περαιτέρω και να το ενισχύσουμε βεβαίω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλει αναφέρουσα για να κλείσουμε τη συζήτηση να πάρει και πάλι το λόγο, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας, ευχαριστώ και την Κομισιόν για τη δουλειά που έχει κάνει για το θέμα αυτό. Επαναλαμβάνω, εμείς θα θέλαμε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μελετήσει το θέμα αυτό κυρίως το θέμα του ε, πεδίου εφαρμογή της ε, απαγόρευσης για, για τις δοκιμές. Το πεδίο εφαρμογή πρέπει να μην είναι τόσο αυστηρό έτσι ώστε να μειωθεί η πρόθεση του Κοινοβουλίου να, να απαγορεύσει τις, ε, τις δοκιμές σε ζώα των συστατικών, τόσο, τόσο λίγων συστατικών που τελικά να γίνει ένα κενό γράμμα αυτή η απαγόρευση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και τις εταιρείες για τις τρίτες χώρες να μην χρησιμοποιούν ε, ζώα για, τα, για, τα, για τις δοκιμές τους. Ε, κυρίως για χώρες όπως η Κίνα και μας στηρίζει σε αυτό και η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι θα διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο σημείο 17. Αναφορά 334 Αναφορά 1236 και αναφορά 1251 του 2011 για την 334 υποθέτω ότι έχετε λάβει όλοι την, το είναι επιστολή του αναφέροντος δεν μπορούν να είναι παρόντες δεν μπορούν να μας παρουσιάσουν την αναφορά τους Νομίζω ότι είναι ο, ο της 1251 ε, εδώ. Θέλετε το λόγο? Thank you. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έρικ Χάτεν ονομάζομαι και είμαι παρόν μαζί με την σύζυγό μου την Ελίζαμπεθ. Η σύζυγός μου και εγώ διευρευνήσαμε τη δυνατότητα να, κάνουμε να πάρουμε τη σύνταξή μας και να πάμε στην έρευνα, στην Κύπρο συγγνώμη, κάνοντας μια έρευνα είδαμε διάφορες εταιρείε ε, ε, για, για, να αγοράσουμε ε, κάποιο, ένα σπίτι. Ε, είδαμε την εταιρεία του κυρίου Κλεάνθου Σάβα, ο οποίος ε, μας είπε ότι ε, χτίζεται μια, ένα συγκρότημα κατοικιών στο χωριό Αναρίτα. Επισκεφθήκαμε τα, τα σπίτια αυτά που πρόκειται να χτιστούν και αποφασίσαμε ποιο θα ήταν το δικό μας οικόπεδο. Γυρίζοντα στο γραφείο, μα πρότειναν ένα πλήρε πακέτο με, με την τράπεζα, με, τους, με συγκεκριμένου δικηγόρου. Μα είπαν ότι είναι αξιόπιστοι. Ο δικηγόρο μα είπαν ότι είναι ο κύριος Γιάννης Παπαζαχαρία, ο οποίος έχει την έδρα του στην Πάφο και πάντα χρησιμοποιεί την Αλφα ε, Bank για, τις, ε, για, τους, ε, για τους πελάτες του. Έγινε μια συνάντηση και με τον Αλφα Bank και με τον δικηγόρο και ο δικηγόρος μας είπε ότι όλα θα πάνε πολύ καλά χρησιμοποιώντας αυτή την τράπεζα γιατί πάντα τον βοηθούσε στις υποθέσεις του. Ε, μας ικανοποίησε η υπηρεσία που μας παρασχέθηκε και του δώσαμε την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσει όλα τα, όλα τα έγγραφα που χρειάζονται. Ε, θεωρήσαμε ότι μπορούμε να τους εμπιστευτούμε τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες ή να ρωτήσουμε περαιτέρω ερωτήσεις. Μα εξηγήσανε βεβαίω για το, το συμβόλαιο. Μα είπαν ότι μπορεί το θέμα τη υποθήκη να είναι πρόβλημα για στην Κύπρο. Ζητήσαμε επίση ε, του τίτλου ιδιοκτησία και μα είπαν ότι το συγκεκριμένο γραφείο ε, δίνει του τίτλου ιδιοκτησία πολύ γρήγορα στου πελάτε του και ότι έχει μια πολύ καλή φήμη και γι' αυτό είναι, πολύ, είναι καλό να, να συνεργαστούμε μαζί του. Μα είπαν ότι μπορεί να κάνει κάποιε έρευνε σε μεταπτυματολόγιο και να ε, και όλο αυτό θα κόστιζε γύρω στα 120 ευρώ. Μα μας είπαν ότι οι δικηγόροι μπορούσαν, μόνο αυτοί μπορούσαν να λάβουν αυτές τις ε, πληροφορίες από το κτηματολόγιο, οπότε τους είπαμε να προχωρήσουν. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει κρεμούσα υποθήκη, οπότε υπέγραψαν ε, εκ μέρους μας το συμβόλαιο. Μετά συνδεθήκαμε με εκπροσώπους της Αλφαβάνκ και μας είπαν ότι η, μόνη συστηνόμενη υποθήκη ήταν μια υποθήκη από Ελβετική Τράπεζα με πολύ χαμηλό επιτόκιο, σε Ελβετικό φράγκο. Μα είπαν ότι έχουν από το γραφείο πάρα πολλού ε, Βρετανού πελάτε και θεωρήσαμε ότι είχαμε, ε, ήταν πολύ καλή η συμφωνία που είχαμε κάνει και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να ε, εμπιστευτούμε τους ανθρώπους αυτούς. Επιστρέψαμε στην ε, Βρετανία και βεβαίως αναμέναμε να έρθει η ώρα για την συνταξιοδότησή μας. Ήρθαμε σε επαφή με τον developer, ο οποίος μας έδειξε και την πρόοδο των κατασκευών. Επίσης μας, ήρθαν σε επαφή μαζί μας πριν από την μετακόμιση μας στην Κύπρο και η τράπεζα και ο δικηγόρος και μας είπαν ότι όλα πάνε καλά. Γυρνώντας στην Κύπρο, ε, είπαμε στον, ε, στο γραφείο ότι, θα, ότι ήρθαμε και πήγαμε στην Αναρίτα για να δούμε το σπίτι. Το σπίτι δεν είχε καμία σχέση όμως με αυτό που μας είχαν στείλει στις φωτογραφίες. Δεν είχε, δεν είχε ολοκληρωθεί τίποτα, μόνο μια γεννήτρια έδινε ρεύμα που βεβαίως δεν ήταν τεράστια για να υποστηρίξει όλες τις ε, κατασκευές, το συγκρότημα αυτό. Η, Ήρθε ένα από το γραφείο και, μας, ε, και του είπαμε ότι είναι διαφορετικό αυτό ε, το οικόπεδο από αυτό που επιλέξαμε. Ε, μα είπαν όμω ότι αυτό είχαμε διαλέξει. Είπαμε να δούμε τον υπεύθυνο, αλλά μα είπε ότι δεν είναι διαθέσιμο και έφυγε. Οπότε δεν είχαμε κανέναν τρόπο εμεί να μπούμε στο σπίτι, κοιτούσαμε από τα παράθυρα γιατί δεν είχαμε κλειδί και είδαμε ότι το, α, και η διαρρύθμιση του σπιτιού δεν, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχαμε διαλέξει. Είχαμε κάνει κάποιε κρατήσει εμεί στο ξενοδοχείο, μείναμε εκεί, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Την επόμενη, φορά πήγαμε στο γραφείο, την επόμενη μέρα πήγαμε στο γραφείο και μα είπαν ότι τα σπίτια που χτίζονται εκεί έπρεπε να χτιστούν με αυτή τη διαρρύθμιση για να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία την Κυπριακή. Και ότι ο developer έχει αγοράσει την, ε, ε, την γη από έναν άλλον developer που είχε χρεοκοπήσει. Μα είπαν ότι ε, κατά λάθο μα είχαν στείλει ε, εκείνε τι ε, φωτογραφίε. Επίση, μα είπαν ότι θα μπορούσαν ίσω να χτιστούν κάπου αλλού ε, σπίτια με το δικό μα με αυτό το σχέδιο που είχαμε επιλέξει και μα είπαν ότι θα μα αναβαθμίσουν μόλις είναι διαθέσιμα τα σπίτια αυτά. Εμεί ήρθαμε σε επαφή με τον δικηγόρο και του είπαμε και μας είπαμε μάλλον ότι θα πρέπει να δεχτούμε την προσφορά που μα γίνεται. Όταν ε, μετακομίσαμε όλα τα σπίτια είχαν τεράστια προβλήματα με ε, βουλωμένου σωλήνες, με πόρτες που δεν έκλειναν, με διαρροές. Ε, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και μας κατηγόρησαν μάλιστα ότι εμείς είχαμε ανοίξει τρύπε στις πόρτες. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα διορθώσουμε τα πράγματα, εγώ δηλαδή αποφάσισα από μόνος μου και ανακάλυψα ότι είχε, είχαν γίνει λαθασμένες συνδέσεις υδραυλικές και βεβαίω όταν φέραμε κάποιου ε, υδραυλικούς το θέμα λύθηκε. Συνέχεια τελείωνε το καύσιμο στη Γιαννήτρια. Είχαμε και προβλήματα τέτοια. Βεβαίω πέρασαν κάποιοι μήνε μέχρι να λυθούν όλα αυτά. Ο developer ποτέ δεν ήρθε σε επαφή μαζί μα, δεν είχε χρόνο για μα. Οπότε θεωρήσαμε ότι αυτό το θέμα έπρεπε να το λύσουμε και να πουλήσουμε την, ε, το σπίτι αυτό. Ακούσαμε μετά κάποιες φήμες ότι ε, ο, ο developer είχε πάρει μια υποθήκη, μια δεύτερη υποθήκη και ζητήσαμε στοιχεία από, το, από, το, από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Πήγαμε λοιπόν στο κτηματολόγιο με τους γείτονές μας και είδαμε ότι έχει ληφθεί η υποθήκη πριν υπογράψουμε εμείς τα συμβολέα μας και ότι αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε λάβει ε, εδώ και ένα χρόνο ως πληροφορίες και μόνοι μας. Δώσαμε τις πληροφορίες αυτές στον ε, δικηγόρο και, το, και αρνήθηκε ότι του είχαμε ζητήσει να πάρει αυτές τις πληροφορίες παρόλο που αυτό είχε γίνει. Μετά από διάφορες έρευνες είδαμε ότι η Alpha Bank έδωσε στον Κλεάνθη Σάβα τη δεύτερη υποθήκη και αυτός δεν πλήρωνε και τώρα χρωστάει περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ κλείσαμε ένα ραντεβού με την Αλφαμπάνκ για να μιλήσουμε με τον, ε, με τον μάνατζερ και ε, αυτοί αρνήθηκαν ότι, ότι υπάρχει κάποια κρίμωσα υποθήκη. Ζητήσαμε να δούμε το τίτλου του ε, γραφείου, έφυγε από το γραφείο και μας είπαν ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν μάθαμε, δεν ήρθε κανένα σε επαφή μαζί μας από την ε, τράπεζα, ούτε από την ε, υπηρεσία για την, ε, από το χρηματολόγιο, ούτε είχαμε πρόσβαση στο φάκελό μας. Μας είπαν ότι έχουν διπλασιαστεί οι πληρωμές, για τις, δόσεις για την υποθήκη μας και θεωρούσαμε ότι ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση είτε να αποπληρώσουμε το δάνειο αυτό, είτε να πάρουμε τίτλους ιδιοκτησίας για το σπίτι μας ο developer μας είπε ότι, ε, ενώ του είπαμε ότι μας είχε εξαπατήσει, αυτός μας είπε ε, ε, είσαι στην Κύπρο τώρα όμως. Εμείς περιμέναμε έξω από το γραφείο του. Το επόμενο πρωί, όταν έφτασε, ζητήσαμε να του μιλήσουμε. Αρνήθηκε να μας δει. Δεν ξέραμε τι ακριβώς να κάνουμε. Γιατί ξέραμε ότι μας είχαν. Νιώθαμε ότι μας είχαν απογοητεύσει όλοι όσοι θεωρούσαμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε. Κάποια από τα προσωπικά μας έγγραφα είχαν ε, κλαπεί, μας ε, απείλησαν κάποιοι έξω από το σπίτι μας. Ε, η, η, τη γυναίκα μου επίσης την χτύπησαν στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, την έριξαν κάτω. Ο μάνατζερ μας είπε να φύγουμε από την Κύπρο και πραγματικά αισθανθήκαμε πάρα πολύ ανασφαλείς και θέλαμε απλώ να παρατήσουμε τα πάντα και να μετακομίσουμε πίσω στη Βρετανία. Είχαμε αγοράσει τρία, τρία ε, σπίτια ε, και δύο αυτοκίνητα γιατί όλα μας τα χρήματα τα είχαμε επενδύσει στην Κύπρο και γυρίσαμε στην, ε, στην Βρετανία άφραγοι. Τώρα ζούμε στο, σε ενοικιασμένο διαμέρισμα. Η υπόθεση στην Κύπρο δεν έχει κλείσει. Τα χρήματα μας τελειώνουν και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά υποθέτουμε ότι απλώς τα πράγματα θα χειροτερεύσουν θα σκεφτόταν κανείς ότι η Αλφα Bank και ο, ο κύριος ε, Γιάννης Παπαζαχαρία θα ήταν αξιόπιστοι και ότι θα μας προστάτευαν από, τα, από τις διάφορες λεπτομέρειες του συμβολέου, το οποίο ο ίδιος υπέγραψε εξ ονόματός μας. Μας ε, εξαπάτησαν, αλλά τελικά βλέπω ότι κανένας δεν διέρευνα την υπόθεση και απλώς αυτοί συνεχίζουν να εξαπατούν τον κόσμο. Προσπαθήσαμε να λάβουμε κάποια συμβουλή από την, ε, στην Αγγλία γι' αυτό, αλλά μας είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι δικηγόροι στην Αγγλία. Είχαμε δύο Κύπριους ε, ε, δικηγόρους που, συνα... που μίλησαν με τους δικηγόρους στην ε, Κύπρο και ούτε αυτοί κατάφεραν να βρουν στοιχεία και δεν μας βοήθησαν καθόλου. Πρόσφατα μας ενημέρωσε ένα δικηγορικό γραφείο ότι η Αλφα Μπάνκ έχει ξεκινήσει μια, ένα δικαστήριο εναντίον μας, το οποίο δεν γνωρίζαμε, στην Κύπρο Μα είπαν ότι έχει στελεί σε μια ε, διεύθυνση στην οποία ποτέ δεν ζούσαμε. Η Alpha Bank πάντα είχε την, το email μας, αλλά δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί μας μέσω email. Απαντήσαμε αμέσως στους ε, δικηγόρους στην Αγγλία και εξηγήσαμε την ε, υπόθεσή μας. Ήρθαν σε επαφή με την Αλφα Bank, η οποία ακόμη δεν τους έχει απαντήσει. Θα δείτε από το συμβόλαιο ότι λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει υποθήκη ούτε για το οικόπεδο ούτε για το κτίριο. Αν ξέραμε ότι υπάρχει υποθήκη για το οικόπεδο δεν θα είχαμε αγοράσει τίποτα προφανώς στην Κύπρο. Μας απογοήτευσε και ο developer και η Αλφαμπάν και ο δικηγόρος. Όλοι έκρυψαν συγκεκριμένα δεδομένα από εμά και συγκεκριμένα στοιχεία η Κύπρος εξακολουθεί έχει να λαμβάνει πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια παρόλο που έχει ε, φερθεί με τέτοιο τρόπο σε Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε και τα λεφτά μας πίσω. Ευχαριστώ. Thank Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσίαση της αναφοράς σας. Από τις τρεις αυτές αναφορές βλέπω ότι δεν είσαστε μόνος σας. Η Κομισιόν η κυρία Ριντού, δεν ξέρω αν έχω προφέρει σωστά το όνομά σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι η Κομισιόν συμμερίζεται τις ε, ανησυχίες του αναφέροντος και των άλλων Ευρωπαίων πολιτών για τη δραματική κατάσταση που αντιμετώπισαν λόγω τέτοιων ε, πρακτικών ε, από τις Κυπριακές Τράπεζες, από δικηγορικές εταιρείες και από τους ε, developers. Η Κομισιόν θα, λάβει όλα τις, ε, θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες δράσεις, στα πλαίσια της εντολής της βεβαίως, για να εξασφαλίσει αποτελεσματική προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και τη σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα ήθελα να σημειώσω παρόλα αυτά ότι σήμερα συζητούμε τρεις αναφορές και θεωρούμε ότι η μία αναφορά η 1236 δεν σχετίζεται με τις άλλες δύο. Αυτή που σας αναφέρω, η 1236, δεν ε, αφορά τον ε, κατασκευαστικό κλάδο. Ήδη έχουμε αναφέρει τι γίνεται με τούτη την ε, με, την, ε, με αυτή την αναφορά, γιατί αυτά τα θέματα άπτονται τη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Δεν μπορεί να παρέμβει η Κομισιόν. Η Κυπριακή Νομοθεσία του 2007, που αναφέρεται εδώ σε τούτη την αναφορά, μεταφέρει τις, ε, την οδηγία για τι αφέμητε εμπορικέ πρακτικέ στο κυπριακό σύστημα και αυτή η οδηγία ε, αφορά θέματα εταιριών προς καταναλωτές. Αυτά για τη 1200 για την 1236 μιλάμε όμως για κάποιους κυβερνητικούς υπαλλήλους που πρέπει να διορθώσουν τις, τα λάθη που έχουν γίνει σε περιπτώσεις αγοράς οικοδομών κτλ. Και μιλούμε για οικοδομές του 2005, δηλαδή πριν την θέση ισχύ. Τη ε, οδηγίας για τις αθέμητε εμπορικές πρακτικές. Οπότε θα επικεντρωθώ μόνο στις άλλες δύο αναφορές που σχετίζονται με την ε, έλλειψη ασφάλειας ε, προς τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει σπίτια στην, στην Κύπρο. Η Κομισιόν σε πολλές περιπτώσεις έχει επαναλάβει ότι η αποτυχία να μεταφερθούν οι τίτλοι δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, αθέμητη εμπορική πρακτική σε κάθε περίπτωση. Γιατί μόνο οι πρακτικές που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της οδηγίας μπορούν να θεωρηθούν αθέμητες αυτές καθ' αυτές. Τούτου λεκθέντος και ε, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, οι εμπορευόμενοι έχουν την υποχρέωση να μην παρέχουν λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που είναι προ πώληση και ε, ζητούνται να παράσχονται πληροφορίες συγκεκριμένε με σαφή, εύληπτο και έγκαιρο τρόπο προς του καταναλωτές. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η έλλειψη αυτών των προσυμβατικών πληροφοριών στους αγοραστές για την, για την ύπαρξη των πιθανών ε, υποθηκών των developers θα μπορούσαν να θεωρηθεί αθέμητη πρακτική για τους σκοπούς της οδηγίας. Οπότε η Κομισιόν θεωρεί ότι ε, η λανθασμένη αναφορά ότι δεν υπάρχει υποθήκη για την προσπόληση, ε, για, προσπό, για την προσπόληση οικοδομή αντίκειται στην οδηγία. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται μόνο σε συναλλαγές που γίνονται μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, δηλαδή μετά το Δεκέμβρη του 2007. Πριν τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, η λανθασμένη μάλλον η, απαγορευόταν η λαθασμένη διαφήμιση από την οδηγία και την παραπλανητική διαφήμιση. Και οι συμβατικοί όροι που δημιουργούν σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δύο μερών προς όφελος της ε, εταιρείας και όχι του καταναλωτή θα έπρεπε να μπουν στις, ε, στην σχετική οδηγία. Εδώ δηλαδή μιλούμε για ε, οδηγία που ισχύει μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση του 2004. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι η βασική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Γι' αυτό η Κομισιόν θεωρεί ότι οι καταναλωτές που είναι θύματα τέτοιων πρακτικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Συνεργασίας ε, Καταναλωτών που υποχρεώνει τις αρχές να διερευνήσουν, να εξεύρουν και να σταματήσουν αυτές τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Στα πλαίσια αυτού του δικτύου οι Βρετανικές ε, αρχές, το, η υπηρεσία για το δίκαιο εμπόριο θα πρέπει να ζητήσουν περαιτέρω ε, έρευνα από τους ε, Κύπριους ομολόγους τους και αν όντως διαπιστωθεί παραβίαση να ζητήσουν την πάυση αυτής της πρακτικής. Επιπλέον, διάφορες πτυχές που σχετίζονται με αθέμητες πρακτικές όπως η αποζημίωση για παραβιάσεις εθνικών συμβάσεων ε, παραμένουν στα χέρια της εθνικής νομοθεσίας και θα πρέπει να να περάσουν στην κρίση των εθνικών δικαστηρίων. Επίσης, η Κομισιόν είναι πολύ ενεργή σε ό,τι αφορά τις ε, ε, τις οικοδομές αυτές ε, ε, και τα δικαιώματα ιδιοκτησία στην Κύπρο. Ήδη έχει ξεκινήσει ένας πολύ αυστηρός διάλογος με τις κυπριακές αρχές και ζητούμε πληροφορίες για τις δράσεις που γίνονται σε εθνικό επίπεδο ώστε να λυθούν τα θέματα πρακτικής και να δούμε τι γίνεται με την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μία από τι βασικέ προτεραιότητε για δράση που αναφέρεται στην ε, έκθεση για την ε, εφαρμογή τη οδηγία ε, για τι αθέμητε πρακτικέ είναι η έναρξη ε, των διαδικασιών επί παραβάση, όπου η Κομισιόν έχει επιβεβαίωση ότι τα κράτη-μέλη δεν συνάδουν, δεν συμμορφώνονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας, μια που αυτό είναι υποχρέωσή τους. Τώρα η Κομισιόν κάνει μια εισβάθους εξέταση των πληροφοριών που έχει λάβει πρόσφατα από τις Κυπριακές Αρχές μετά από ένα δεύτερο αίτημα για ενημέρωση. Και οι υπηρεσίες Κομισιόν θα προωθήσουν ε, και θα συνεχίσουν την μελέτη και θα ξεκινήσουν την ε, διαδικασία επιπαραβάση εάν θεωρήσουμε, ε, έχουμε μάλλον συγκεκριμένα στοιχεία που λένε ότι οι εθνικές αρχές τη Κύπρου δεν μεταφέρουν σωστά και δεν εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλει κάποιο συνάδελφο το λόγο. κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι φίλη της Κύπρου και ε, πάντα ε, είχα πολλές, πολύ στενέ επαφέ και με συναδέλφου και για το θέμα των αγνοωμένων και ζούσα και στην Κύπρο μάλιστα κάποια χρόνια. Όταν εξελέγει το 2009 έλαβα πολλέ ε, αναφορέ από ε, ανθρώπου στην εκλογική μου περιφέρεια που είχαν επενδύσει σε περιουσία στην Κύπρο. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο Χριστόφια τον απερχόμενο για το θέμα αυτό και διάβασα την αναφορά που λέει ότι υπάρχει ένα στοιχείο ε, σε αυτές τις διαδικασίες. Εγώ θα ζητούσα από την Επιτροπή μας, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν δαπανίσει όλο αυτό το χρόνο και έχουν κάνει τόση προσπάθεια να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο και θεωρούν ότι δεν τους ακούει κανείς ή τους, ε, δεν τους καταλαβαίνουμε, νομίζω ότι είναι ε, χρέος της Επιτροπής μας να κάνει ένα βήμα πίσω, να ακούσει και να δει τι έχει παρεξηγήσει. Οπότε υποστηρίζω απόλυτα το να αναβάλουμε το θέμα αυτό και να μας δώσουν οι αναφέροντες περισσότερες πληροφορίες. Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό για την Κυπριακή κυβέρνηση. Οι Κύπροι υποστηρίζουν απόλυτα την ε, ένταξή τους στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, των τελευταίων συμβάντων εξαιρουμένων. Έχουν, θεωρούν ότι έχουν κερδίσει από την ένταξή τους στην Ένωση και έχουν ωφεληθεί. Βεβαίως με τα ωφέλη αυτά έρχονται μαζί και κάποιε ευθύνε. Μπορώ να καταλάβω ότι ίσως να θεωρούν ότι ε, αυτοί είναι ξένοι που αγοράζουν τη γη μας. Εντάξει, ως εκεί ναι, αλλά έχουν ε, μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνε που έρχονται μαζί με αυτό. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί. οι αναφέροντες έχουν κάνει πολλά, πάρα πολλά και πιστεύω ότι είναι δική μας η ευθύνη τώρα, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Το πρώτο θέμα είναι να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι ε, αναφορές και θεωρώ ότι η Κομισιόν πρέπει να είναι πιο ενεργή σε αυτή την ε, φάση. Αν όντω βρείτε αν κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, νομίζω ότι σίγουρα θα βρείτε στοιχεία για να υποστηρίξετε τους, α, ε, ε, τους αναφέροντες. Δεν μπορεί να πρέπει να κάνουν αυτοί όλη τη δουλειά της απόδειξης α, ε, της απάτης. Δεν ξέρω αν θέλει ο αναφέρον να πάρει και πάλι το λόγο. Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι προσπαθούμε να πάρουμε τη γη των Κυπρίων. αυτοί έρχονται στις χώρες μας και προσπαθούν να πουλήσουν αυτή την ε, γη και προσπαθούν να εξαπατήσουν άλλους ανθρώπους όπως εξαπάτησαν και εμάς. Γι' αυτό ε, ζητώ πραγματικά τη βοήθειά σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Να είστε σίγουροι ότι θα έχετε τη στήριξή μας. Ελπίζουμε να υπάρξει επιτυχής κατάληξη. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή στην εμερήσια διάταξη. Ζητώ την κατανόησή σας ε, λόγω ανωτέρας βίας. Πρέπει να δούμε το σημείο 16, την αναφορά 336 του 2012, τώρα και μετά θα πάμε στο σημείο 18 για τις κοινωνικές υποθέσεις. Ζητώ την κατανόησή σας. Οι αναφέροντες της 336 ε, νομίζω ότι είναι εδώ Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρίε και κύριοι. Μπριγκίτε Ντάμ ονομάζομαι και είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρου τη Δισλανδική Εταιρεία Προστασία των Ζώων για τη συστηματική κοπή τη ουρά των χειριδίων. Είναι τεράστιο το στρες που προκαλείται στα χειρίδια η οδηγία για το Συμβούλιο ε, ορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ε, χειριδίων και λέει ότι η κοπή της ουράς δεν πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πριν από την ε, κοπή της ουράς θα πρέπει να λαμβάνονται άλλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη και το, την, τα αποθέματα, τα, τα, τα κοπάδια, τον αριθμό των κοπαδιών και των περιβάλλων οι αριθμοί δείχνουν ότι γίνεται συστηματικά η κοπή ε, της ουράς των χειριδίων και δεν έχουν ληφθεί κα, ε, απαραίτητα, τα απαραίτητα μέτρα από τις δανέζικες αρχές. Αυτό επιβεβαιώθηκε από μία έναν έλεγχο στην ε, Δανία το 2010 από την Κομισιόν. Η, ο έλεγχος λέει, και παραθέτω, η κοπή της ουράς των χειριδίων γίνεται συστηματικά χωρίς επαρκή διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές εάν έχουν γίνει προσπάθειες από τον ε, κτηνοτρόφο να βελτιώσει τις ε, περιβαλλοντικές συνθήκες ή το σύστημα διαχείρισης. Από τότε ούτε η παραγωγή χειριδίων ούτε οι αρχές της Δανίας έχουν κάνει κάποια αλλαγή στις πρακτικές τους και συνεχίζουν να, ε, αυτή την πρακτική. Το 2011 Εμεί, η Δανέζικη Εταιρεία Προστασία των Ζώων, υποβάλαμε προσφυγή στην Κομισιόν, γιατί η κοπή τη ουράς των χειριδίων ε, γίνεται και σε άλλα κράτη-μέλη. Υπήρχαν προσφυγέ από τη Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Και αυτό το θέμα είναι ευρωπαϊκό. Στην απάντησή μα στην προσφυγή, η Κομισιόν αναγνωρίζει το πρόβλημα έτσι όπω το έχουμε περιγράψει και επιβεβαιώνει παρόμοιε πρακτικέ και σε άλλα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν δεν θα ξεκινήσει τη διαδικασία παραβάση παρόλα αυτά, αλλά όπως και προηγούμενα χρόνια θα συνεχίσει να εμπιστεύεται την επικοινωνία μεταξύ των διαφορών μερών και την ε, ε, ενημέρωση που υπάρχει. Αυτό θεωρούμε ότι είναι απογοητευτικό. Ε, όπως, είναι, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη και οι δανέζικες αρχές και η βιομηχανία γνωρίζουν απόλυτα την νομοθεσία και πώς μπορούν όλα αυτά να αποτραπούν. Αλλά χρειάζονται περαιτέρω πόροι κυρίως εξοπλισμός και ε, χώρος, ε, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις για, τις, για τα χειρίδια. Επίσης ε, είναι δύσκολο να καταγραφούν τα στοιχεία γιατί τα προβλήματα της κοπής της ουράς των χειριδίων γίνονται μόνο όταν τα ζώα πηγαίνουν προσφαγή. φαγή. Επομένως δεν μπορούν να υπάρξουν τα στοιχεία ήδη από πριν η πρακτική αυτή είναι προληπτική και δυστυχώς καμιά ενημέρωση δεν μπορεί να αλλάξει μια τέτοια πρακτική. Τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να κόβουν τις ουσουρά των χειριδίων, αν και υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Λιθουανία, η Σιουηδία που συνάδουν με τις, και συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας. Είναι λοιπόν σαφές ότι τα κράτη-μέλη που συμμορφώνονται έχουν προφανώς περισσότερους πόρους για να το κάνουν αυτό η ε, παραγωγή ας πούμε στην ε, Γερμανία ε, έχουν εισάγει 9 εκατομμύρια χειρίδια προσπάχυνση από τη Δανία. Οι Γερμανοί κτηνοτρόφοι θέλουν να αγοράσουν τέτοια χειρίδια. Επομένως, χώρες που συμμορφώνονται δεν έχουν χειρίδια χωρίς ουρά για να πουλήσουν και επομένως δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά. Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίε επί παραβάση. Παρ' όλα αυτά, αυτό το έχει αρνηθεί επανειλημμένα η Κομισιόν. Εμεί θέλουμε να κάνουμε άλλη μία πρόταση για το πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην οδηγία, να, να, να μεταβεβαστεί το βάρος της απόδειξης στους ε, κτηνοτρόφους ε, ε, των χείρων προς σφαγή. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να λέει ότι καμία εκμετάλλευση που σφάζει χειρίδια δεν θα πρέπει να δέχεται χειρίδια με, κομμένη ουρά εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι αυτό έγινε ε, λόγω συγκεκριμένων, μετά από συγκεκριμένες μάλλον προϋποθέσεις. Η κοπή τη ουρά πρέπει να είναι το τελευταίο, η τελευταία λύση. Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, ασυνέπειε με την, ε, με την ε, διατύπωση οδηγία. Θα πρέπει η οδηγία να εφαρμοστεί και να είναι πιο εύληπτη. Επίσης, προτείνουμε να υπάρχει δήλωση από κτηνίατρο μαζί με, την, με τα συνοδευτικά έγγραφα που θα λέει ότι σε αυτή την ε, συγκεκριμένη εκμετάλλευση έχουν υπάρξει προβλήματα κοπής τη ουράς των χειριδίων και δεν υπήρξε, πρόβλημα, δεν υπήρξε δυνατότητα να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτή η, λύση, αυτή η αναφορά θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά και θα πρέπει να υπάρξουν και δράσει για να λύσουμε την ε, κατάσταση αυτή. Οι αρχές μετά θα πρέπει να απαιτήσουν να δούνε την εκτινετική αυτή δήλωση όταν ελέγχουν τις εκμεταλλεύσεις. Και είναι βεβαίω πολύ σημαντικό αυτό το προφανές κενό μεταξύ της, ε, των απαιτήσεων της οδηγίας και της ε, πραγματικότητας να κλείσει. Αυτό πρέπει να γίνει για να εξασφαλίσουμε την ευζοία των χειριδίων που, τα οποία θέλει να προστατεύσει η οδηγία, αλλά και να εξασφαλίσουμε την, το σεβασμό της, ε, της νομοθεσίας που έχει δημοκρατικά αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντας, το σημείο αυτό είναι ένα, θέμα στο οποίο υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές. Δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα λοιπόν από αυτού. Η Επιτροπή έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Όντως το πρόβλημα είναι ευραία, ε, σε μεγάλη κλίμακα. Η Επιτροπή όμως δεν θεωρεί ότι υπάρξουν αλλαγή των κανόνων αλλά αυτό που χρειάζεται είναι μία κατάρτιση, ενημέρωση. Υπάρχουν πολλά μέτρα που έχουν ληφθεί. Το πρόβλημα της κοπής της ουράς είναι περίπλοκο, όπως τα ανέφερε και η προαλήσασα. Σε χώρες όπου που ε, εκτρέφουν χειρίδια εφαρμόζουν την απαγόρευση αυτή διότι πια έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά οι Ολλανδοί και οι Δανείοι που κάνουν εξαγωγές σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτές τις χώρες να έχουν την απαγόρευση αυτή διότι διότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα άμα κανείς κόψει την ουρά. ε, για παράδειγμα καμιά φορά όταν πλήττουν τα γερίδια έχουν την τάση τα μένα δαγκώνουν την ουρά του, των άλλων. Επίσης υπάρχουν ομάδες που είναι μικτές ε, τα ζώα τα οποία συγχροντίζονται με άλλα ζώα μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα. Μετά υπάρχει το έδαφος, η ποιότητα του αέρα, ε, πολλές στοιχές δηλαδή σε σχέση τώρα με όλα αυτά, η φιλοδοξία της Επιτροπής είναι καταρχήν να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές. Η στρατηγική που εγκρίθηκε πέρσι για το ευζήν των ζώων οδηγούσε σε μια σειρά βέλτιστων πρακτικών που θα τις έχουμε την επόμενη χρονιά και θα υπάρξει οδηγία για τα για τους χείρους. Φέτος όμως είχαμε την προτεραιότητα να δούμε το θέμα που έχει να κάνει με την, ε, τις ομάδες ζών. Γίνεται τώρα έργο πάνω σε αυτό. Εδώ και λίγο καιρό ξεκινήσαμε και του χρόνου θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Όντως, όταν υπάρχει γενικό πρόβλημα, το, το θέμα, η προσέγγιση των κυρίων δεν είναι η επιτυχούσα προσέγγιση. Ε, είναι ενδιαφέρουσες προτάσεις που, που γίνανε, αλλά δεν θα αντιμετωπιστεί ίσως έτσι το τεχνικό πρόβλημα, διότι είναι ένα τεχνικό πρόβλημα. Επίσης, μετά από αυτό το, την αναφορά κάναμε επαφή με αρχές στη Δανία και είδαμε ότι υπάρχουν πολλές ε, παραβάσεις. Και κοιτάμε να, τους, να ενταχθούν ε, εκεί οι αρχές στις κατευθυντήρες γραμμές. Και θα κλείσω σε μια γενική παρατήρηση που έχει να κάνει με, το, με τις καλές συνθήκες για τα ζώα. Η Επιτροπή θέλει να προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου, κάποια κέντρα δηλαδή αναφοράς, που... και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υποστήριξε είναι λοιπόν μία από τις προτάσεις που θέλουμε να προχωρήσουμε. Είναι, υπάρχει τέτοια ανάγκη. Δηλαδή όχι μόνο νομοθεσία αλλά τεχνικά μέτρα στις χώρες μέλη να γίνουν καταλύτερα κατονητές οι, οι πρακτικές που πρέπει να υπάρχουν και να εφαρμοστούν σωστά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Συνάδελφε Τέιλορ, θέλεις το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την αναφέρουσα και ευχαριστώ και την Κομισιόν για την απάντησή τη. Δεν είναι μόνο δανέζικο πρόβλημα αυτό. Ε, είναι σύνηθε φαινόμενο στη Γαλλία και στη Γερμανία η κοπή τη ουρά των χειριδίων. Απ' την άλλη, κάποιε χώρε όπω η Σουηδία και η Φιλανδία και η Λιθουανία δεν κόβουν τι ουρέ των χειριδίων. Αυτή η πρακτική είναι θέμα ευζοία. Ε, έχει να κάνει και με την ε, πυκνότητα των ε, κοπαδιών και με το χώρο που έχουν τα χειρίδια και βεβαίως και με την αποφυγή του στρες κατά την όλη διαδικασία κοπής. Είναι σαφές λοιπόν ότι η Κομισιόν αυτό που κάνει δεν πετυχαίνει έτσι ώστε να αποτρέψει αυτή τη συστηματική κόπη της ουράς των χειριδίων. 99,2% όλων των χειριδίων στη Δανία ε, έχουν, τους έχουν κόψει τις ουρές. Οπότε οτιδήποτε κάνει η Κομισιόν δυστυχώς δεν πετυχαίνει. Και σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ζητήσουμε διαδικασία επί παραβάση. Είναι δύσκολο βεβαίως να ακολουθηθεί η οδηγία γιατί οι κτηνοτρόφοι των χειριδίων ε, τα πουλούν σε εταιρείε πάχυνση. Ίσως και σε τρίτες χώρες κάποιες φορές. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πριν την πώληση τα... γίνεται συστηματική κοπή της ε, ουράς των χειριδίων. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε την νομοθεσία και είναι ε, ενδιαφέρουσες οι προτάσεις που γίνονται, αλλά πρέπει να μπορούμε και να αιτιολογήσουμε και να αποδείξουμε ότι χρειάζεται, χρειάζεται και είναι αιτιολογημένο η συστηματική κοπή της ουράς και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το επιστοποιήσει η κτηνίατρος. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν, η θέση μάλλον της Κομισιόν δεν είναι αποδεκτή. Συμφωνώ ότι η διαδικασία παραβάση θα πρέπει να ξεκινήσει και δεν αρκεί απλώς να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον, να ελπίζουμε ότι το καθεστώς αυτό θα, αυτό λειτουργήσει. Πρέπει να προχωρήσουμε και σε πράξεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Μάργαρετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θυμάμαι ότι και στην ε, ομάδα για την ευζοία των ζώων στην Ίντε είχαμε μια μακρά παρουσίαση για την ε, πρακτική αυτή και ήταν και λίγο... Ε, μας έφερε σε δύσκολη θέση το γεγονός ότι μια τόσο σαφής νομοθεσία παραβιάζεται. Για χρόνια το βλέπουμε και είναι, είναι περίεργο που η Κομισιόν δεν κάνει κάτι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Οι κτηνοτρόφοι χειριδίων θέλουν να έχουν ευζοία για τα, για τα ζώα τους, αλλά δεν έχουν καμία τύχη στην αγορά, γιατί επιτρέπουμε εμείς ακόμα αυτή την, α, αυτή την πρακτική. Ξέρετε, Κομισιόν, και εσείς και εγώ το ξέρουμε, ότι είναι ένα σαφές μήνυμα αυτή η πρακτική της κοπής της ουράς των χειριδίων, ότι δεν έχουν καμία καλή μεταχείριση, γιατί είναι κάτι που γίνεται συστηματικά. Νομίζω λοιπόν ότι η, Κομισιόν δεν θα πρέπει να μας απαντάει ενημερώστε τους κτηνοτρόφους, εσάς παρακαλώ. Αυτοί που θέλουν να ενημερωθούν, θα ενημερωθούν. Η Κομισιόν πρέπει να επιμείνει στην τήρηση της νομοθεσίας. Αυτό είναι το δικό σας το καθήκον, αυτή είναι η δουλειά σας. Να εξασφαλίσετε ότι θα εφαρμοστεί η νομοθεσία. Επομένως, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέσα στα χέρια μας, όχι μόνο ωραία λόγια. Η πρότασή σας να συνδέεται ε, ε, η τεκμηρίωση με τα ε, με τις εκμεταλλεύσεις που έχουν το πρόβλημα δεν είναι τα χειρίδια που έχουν το πρόβλημα είναι τα μεγάλα, οι μεγάλοι χείροι που έχουν το πρόβλημα είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τα ζώα πάχυνση οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να την αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή και να θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στην Κομισιόν τι θα κάνει ώστε να είναι σαφής η εφαρμογή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε και την αναφέρουσα που μας παρουσίασε την ε, αναφορά. Θα πρότεινα βεβαίως να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, βεβαίως να θέσουμε τα ερωτήματα στην Κομισιόν, βεβαίως να ε, ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να ξεκινήσει τη διαδικασία παραβάση και να είναι πολύ πιο αυστηρή, γιατί σίγουρα η Κομισιόν κατάλαβε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερω ικανοποιημένοι με την, απο... με την απάντηση που μας δόθηκε. Θέλω να πιστεύω. Ένα σχόλιο. Έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή χειριδίων στην ε, Δανία. Αλλά το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται στη Δανία. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε ποιε είναι οι χώρε όπου γίνονται αυτέ οι πρακτικοί, οι κάτω η Γερμανία, όποιε και αν είναι. Και, σε, και προ αυτέ να στραφούμε, όχι μόνο στη Δανία. Η πρόεδρο χωρί μικρόφωνο. Let me thank you to the petitioner. Ωραία. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν την αναφέρουσα μας παρουσίασε και την αναφορά και το πρόβλημα που υπάρχει, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 18. Αναφορά στα πλαίσια των κοινωνικών υποθέσεων. Αρκετές αναφορές έχουμε εδώ. Η αναφορά 267, 474, 479, 483, 625, 762, 1144, 1261. Όλες από πέρσι. Να δώσω αμέσως τον λόγο στον κύριο Κούτη. Είναι παρόν. Ωραία. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, Λάσλο Κούτι και είμαι πρόεδρος για την Ένωση Υπεράσπιση των Συμφερόντων το, με, Ένωσης με 10.000 μέλη για τα συμφέροντα των ατόπων που λαμβάνουν πρόεδρες στην δεξότηση. Ε, και θέλω να σας πω σχετικά με την κατάσταση του καθεστώτος πρόεδρος στην στην Ουγγαρία. Να σας πω ότι κάθε κράνος μέλος έχει δικαίωμα βέβαια να αλλάξει όπως επιθυμεί το πρόγραμμα κοινωνικής του ασφάλισης. Αλλά δεν είναι αυτό που έγινε στην Ουγγαρία. Είδου τι έγινε. Την 1η Ιανουαρίου του 2012 τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος που αφορούσε εκείνους που έτσι και αλλιώς εδώ και 10 χρόνια ήταν συνταξιούχοι και τους αφαίρεσε την ιδιότητα την ιδιότητα συνταξιοδοτημένου ατόμου. Δεν ήταν μόνο από αστυνομικά σώματα ή στρατιωτικά σώματα, ήταν ε, και από γιατρούς, ήταν από οδηγού, ήταν, ήταν από κόσμο και κόσμο. Και ας πούμε, να σας πω για όσους εργάζονται σε, στον τομέα της ακτινογραφίας, και ακριβώ λόγω της ακτινοβολίας έπρεπε να αποσυρθούν. Από την άλλη μεριά όμω τους ζήτησαν περαιτέρω χρόνια ε, υπηρεσίας και ακόμα και μέλη των αστυνομικών σωμάτων που ε, έκαναν υπερορίες Πάσχα, Χριστούγεννα, ε, νέο έτος και δεν τους έδιναν καμία αμοιβή. Και όπως είχαν δικαίωμα πάντως πήραν την σύνταξή τους και εγώ έλαβα τη σύνταξή μου ε, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που υπήρχε, το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τώρα μου αφαίρεσε αυτό το δικαίωμα το κράτος καιρό μετά. Δεν έχω πια το δικαίωμα να λαμβάνω τη σύνταξή μου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή σαν να αγοράζω ένα καρβέλι ψωμί και μετά να μου πούν το ψωμί που αγόρασες δεν είναι δικό σου». Δεν είναι ότι θέλω το παντεσπάνι μου, θέλω ένα ψωμάκι, δεν ε, το θέλω πολυτελείας, αλλά μου το αφαιρούν. Και εδώ θέλουμε να δούμε ακριβώς αυτό το καθεστώς, το, αυτή είναι δηλαδή την κεκτημένη ε, του, των συνταξιωμένων ατόμων. Δεν ισχύει πια. Είναι κόσμος που είχε ήδη συνταξιδοτηθεί νόμιμα και τώρα δεν μπορούν να έχουν πια σύνταξη και μάλιστα αναδρομικά ισχύει αυτό. Και θεωρούμε ότι είναι, δεν μπορεί να συνδυαστεί αυτό, δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εντάξει, ο κ. Μπαρόζο, ο πρόεδρος της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποίησε την κυβέρνησή μας ότι θα έπρεπε να σεβαστεί η κυβέρνησή μας τις δημοκρατικές αξίες. Συμφωνούμε με τον κύριο Μπαρόζο, πιστεύουμε θα πρέπει να μην παραβιάζονται αυτές οι δημοκρατικές αξίες και αρχές. Λοιπόν, με το σχέδιο αυτού νόμου να σας πω ότι η κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε διάλογο με κανέναν από τους συνταξιούχους. Από την άλλη μεριά βέβαια συζήτησε με τους δικάτα των εργαζομένων. Άλλοι όμως είναι αυτοί. Λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, μην ξεχνάμε και τον αναδρομικό χαρακτήρα των μέτρων. Βλέπουμε ότι εξαφανίζεται η σύνταξη αυτών των ατόμων και κόσμος που εδώ και δέκα χρόνια λαμβάνει σύνταξη τώρα τους αφαιρούν το δικαίωμά τους. Θα πρέπει να αλλάξουν εντελώς τη ζωή τους και ο νόμος 107 του 2011 αυτό θεσπίζει. Σας ευχαριστούμε. Μας παρουσιάσετε την ε, αναφορά. Ζητώ συγγνώμη αν ε, προφέρω λάθος τα, τα ονόματά σας, αλλά δεν μιλώ ουγγρικά. Ο δεύτερος αναφέρον που θέλει το λόγο είναι ο κύριος Κάτους. Ελπίζω ότι το λέω σωστά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάρο Εκατούς. Είμαι από την Ουγγαρία. Εκπροσωπώ 3.000 άτομα. 1.800 άτομα υπογράψανε το 1860 συγκεκριμένα το, την αναφορά που έχετε μπροστά σας θεωρώ ότι είχα μεγάλη τύχη το να συμμετέσχω στο, στο ε- έργο των τελωνιακών όταν ενετάχθη η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορώ να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή στην Ουγγαρία δεν μπορώ να ασκήσω ένα τέτοιο δικαίωμα και έρχομαι εδώ στη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνω. Και οι σύντροφοι που με ακούνε τώρα στην Ουγγαρία και ελπίζουν ότι ε, εδώ στις Βρυξέλλες στο κέντρο της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια βοήθεια και ελπίζουν και εύχονται, προσεύχονται μάλιστα να εισακουστεί αυτό τους, αυτή τους η αναφορά. Και ότι δεν μπορεί να υπάρχουν νόμοι με αναδρομική ισχύ. Άτομα που δουλέψαν 25 ή πιο πολύ και είχαν μια δραστηριότητα στα πλαίσια πάντοτε διαταγμάτων και εθνικών νόμων να βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη ε, άτομα χωρίς δικαιώματα. Μιλάμε για 43.000 τουλάχιστον άτομα από, από τη μια στην λοιπόν όλα αυτά τα άτομα βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου λόγω του, της, ενός νόμου εδώ και 1,5 χρόνο το άλλαξε η κατάστασή τους και υπάρχει μάλιστα και αναδραμική ισχύ σε αυτό το νόμο. Και καταλήγουν άλλα άτομα τα οποία ε, έχουν την ελάχιστη θα λέγαμε ε, αποζημίωση. και καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους. Το 1947 στον παππού μου αφαιρέσανε το δικαίωμα του ε, στη σύνταξη όπως κάνουν τώρα σε μένα. Και ο άνθρωπος μετά από αυτά τα γεγονότα πέθανε και γρήγορα γρήγορα. ένα, μια χώρα μέλος να ανοίξει, να αλλάξει τους νόμους και να αλλάξει τα δικαιώματα ενός εργαζομένου με αυτόν τον τρόπο, και έχουμε να κάνουμε άτομα τα οποία έχουν δεχθεί αυτές τις αλλαγές έχουμε να κάνουμε άτομα τα οποία υπεραμεινθήκαν τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αγωνιστήκαν για δημοκρατικέ αρχέ. Το θέμα λοιπόν τίθεται. Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στις λίγε σελίδε που είναι η απάντησή τη, ε, να κλείσει έτσι ένα θέμα. Ελπίζουμε να επανεξετάσουν το θέμα υπάρχει αρχή τομή διάκριση που πρέπει να γίνει σεβαστή και επίση να πω έχουμε ε, να κάνουμε άτομα τα οποία είχαν υψηλή προστασία και σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτά, τα άτομα σήμερα χάνουν 16% της συνταξή του χωρίς να ξέρουμε γιατί. Μπορεί κανεί να έχει νόμισμα αναδρομική ισχύ. Εγώ είμαι Ούγγρος πολίτης, δούλεψα 25 χρόνια, έκανα όλη αυτή τη διαδρομή στο Στρασβούργο και στην Επιτροπή και θεωρώ αναξιοπρεπές αυτό. Μπορεί κάποιοι να πούνε ότι αυτό είναι μια υπόθεση καθαρά ογκρική. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Αλλά τότε ναι, δεν λαμβάνουμε υπόψη τις ιστορικά γεγονότα που οδηγήσαν στη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία ενός ειρηνικού χώρου στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να διγενεχτούμε κάτι τέτοιο στη Βουδαπέστη. Ο Φραγκίσκος ο πρώτος, ο Πάπας, είπε το εξή στην Αργεντινή. Οι νόμοι και το Σύνταγμα έχουν δημιουργηθεί για να τα σεβόμαστε και όχι για να τα αλλάζουμε όποτε μας καπνίσει. Εδώ και ένα μισή χρόνο τολμήσαν να αλλάξουν το σύνταγμα στην Ουγγαρία για να μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο με τις ε, συντάξεις είναι απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει στηρίζει σε καμία βάση που, με ένα θεμελιώδες δικαιώμα τα άτομα τα οποία έχουν ε, θεσπίσει τέτοιου νόπου και ελπίζουν να μην κοιτάζουν τώρα να σκεφτούν το εξώ. Οι αστυνομικοί, άλλοι ε, άτομα τα οποία φτάνουν στην ηλικία των 64 χρόνων. Οι, ε, ε, ε, οι στατιστικές δείχνουν αντιθέτως εμείς πρόκειται να, να πεθάνουμε νωρίτερα. έχω πάει σε τουλάχιστον σε καμιά πενταριά κηδείες παλιών συναδέφων. Γιατί λοιπόν, γιατί δεν καταλάβανε στη Βουδαπέστη ότι υπάρχει αυτό το δικαίωμα και τι έχουν κάνει, μας αφαιρούν αυτό το δικαίωμα. Πώς μπορεί κανείς να αφήσει ένα πυροσβέστη σε μεγάλη ηλικία να δουλεύει. Πώς μπορεί να το περιμένει κάνει κανείς αυτό. Ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα. Το παλιό σύστημα συντάξεων ίσως να μην ήταν βιώσιμο Καλά, καταλαβαίνω, μίλησα με πολύ έτσι ε, συναισθηματική φόρτιση. Ελπίζω να επιστρέψουμε στη χώρα μας με τη δική σας ε, υποστήριξη. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας. Ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, δεν ε, χρειάζεται να απολογίσετε. Την κυρία Χέλγα την κυρία Πόπελμαν να ακούσουμε από την Κομισιόν να μας απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που δίνετε στην Κομισιόν την ευκαιρία να απαντήσει σε αυτές τις έξι αναφορές που υπευλήθησαν στην Επιτροπή σας από Ούγγρους πολίτες. Αν μου επιτρέπετε, θα απαντήσω σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά το τι δεν μπορούμε να κάνουμε και γιατί. Και το δεύτερο θα αφορά τα όσα μπορούμε να κάνουμε, ήδη κάνουμε και γιατί τους ακούμε με μεγάλη προσοχή. Οι αναφορές, οι έξι αυτές αναφορές αφορούν ένα πακέτο μεταρρυθμιστικό για τις συντάξεις στην Ουγγαρία που υιοθετήθηκε πέρσι. Ήδη είδαμε ένα θέμα που εμπίπτει στον ίδιο τομέα που ήταν στο σημείο 9 της ημερής διάταξης σήμερα που πάλι αφορά το πακέτο αυτό το μεταρρυθμιστικό της Ουγγαρίας. Τώρα εδώ έχουμε αναφορές που περιλαμβάνουν 2866, ε, που συμπεριλαμβάνουν 2866 υπογραφές. Και βεβαίως ε, περιλαμβάνουν και τις ανησυχίες μιας ε, ομάδας δημοσίων υπαλλήλων για την, για την κατάργηση της πρόορης συνταξιοδότησης συνοριοφυλάκων και αστυνομικών που ήδη έχουν κατοχυρώσει εξωτερικά δικαιώματα με συγκεκριμένα κοινωνικά επιδόματα. Κατανοώ και εγώ και οι συναδελφοί μου ότι κυρίως για ανθρώπους που έχουν εργαστεί σε αυτούς τους πατριωτικούς κλάδους, αν μπορώ να το πω έτσι, στρατιωτική υπηρεσία, αστυνομική, ε, υπάρχει και ένα αίσθημα περηφάνειας. όταν βλέπεις ότι τα συνταξιδοτικά σου δικαιώματα μεταφράζονται σε κάποια ελάχιστα κοινωνικά επιδόματα, ε, προφανώς η περηφάνεια σου πλήττεται. Γνωρίζω την κατάσταση και την ε, κατανοώ πλήρως. Έχετε δει βεβαίως και τις επίσημες απαντήσεις μας, οπότε πρέπει να σας επαναλάβω το πώς έχει η κατάσταση νομικά. Ο σχεδιασμός των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης γενικώ είναι σχεδόν στην απόλυτη αποκλειστικότητα των κρατών μελών. Αυτό αναφέρεται ρητά στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το, σύνταγμά μας ουσιαστικά, είναι και το δικό σας σύνταγμα πια ως μέλη της Ένωσης Ουγγαρία. Οι αναφέροντες λένε ότι η νομική πράξη της Ουγγαρίας υπονομεύει αυτή την κατάσταση για, την, α, για τους αστυνομικού για τους αστυνομικούς κτλ. και ότι παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να μπορούσε να, υπο, να ε, ε, ορίσει το πώς θα, κάνει, πώς θα διαρθρώσει το, κοινωνικό, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης η Ουγγαρία. Βεβαίως μιλήσατε και για τη θέση ισχύ αυτής της ε, μεταβατικής περίοδου. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα λόγο στο πώς θα οργανώσετε εσείς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισής σας. Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να παρέμβουμε. Ε, δεν γίνεται να υπάρξει δηλαδή ευρωπαϊκή παρέμβαση για να ακυρώσουμε το, το σχέδιο της ε, κυβέρνησής σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ως προς αυτό. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε καθόλου. Γιατί προφανώς θα υπάρξει λαϊκή ε, κινητοποίηση. Στην επίσημη λοιπόν απάντηση που έχουμε δώσει και αναφέρεται στις έξι αυτές αναφορές μιλά για τα κράτη-μέλη που αφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, δεν ε, υπάρχει άμεση παρέμβαση. Και βεβαίως για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης δεν ε, υπάρχει κανένα θέμα. Η Κομισιόν λοιπόν δεν μπορεί να δώσει οποιαδήποτε άλλη απάντηση, ας πούμε να ξεκινήσει η διαδικασία η παραβάση. Δεν, έχουν, δεν έχουμε αρμοδιότητα τέτοια και ούτε μέσα για να το πράξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διακριτική μεταχείριση, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να πάει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και φαντάζομαι ότι θα το, θα το πράξετε. Δεν ξέρω βέβαια για το κατά πόσο θα είναι παραδεκτό αλλά εκεί θα λάβετε και νομική απάντηση. Αυτά λοιπόν για το, πώς, ε, για, το, ε, για, το κομμάτι που αφορά το τι δεν μπορεί να γίνει από νομική πλευρά. Πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά τις ε, δράσεις της Κομισιόν με τα κράτη-μέλη. Μιλούμε για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, για το σχετικό πλαίσιο από την ε, οικονομική κρίση που χτύπησε όλα τα κράτη-μέλη πολύ σκληρά, τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Κομισιόν και μετά από ενθάρρυνση της Κομισιόν έχουν εκπονήσει κάποια εργαλεία, κάποια μέσα, τα οποία έχουν αρχίσει πια να δημιουργούν και ένα ορόσημο το οποίο μας ε, εκπλήσει και εμάς η Κομισιόν χρόνια ε, προσευχόταν, παρακαλούσε να υπάρξει μια τέτοια ενεργή απάντηση από τα κράτη-μέλη και τώρα υπάρχει. Αυτό είναι το βήμα στο οποίο θα συζητηθεί και η ερώτησή σας. Έχουμε την ε, Ευρώπη 2020, έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όπου τα κράτη-μέλη υποβάλλουν ε, στην ε, Κομισιόν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα. Το επόμενο το περιμένουμε τον Απρίλιο, τον επόμενο μήνα δηλαδή. Και η Κομισιόν προτείνει στο Συμβούλιο ποια γραμμή να, να πάρει για, αυτές τις, ε, για αυτά τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα. και δίνει και τη γνώμη της για την εφαρμογή, καθώς επίσης και για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες. Γιατί βλέπουμε ποιε είναι οι κοινωνικέ επιπτώσει τη της οικονομική κρίση. Δεν θέλω τώρα να ε, μπω σε λεπτομέρειε, γιατί εσεί σας ενδιαφέρει αυτό το ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά θέλω να πω απλώ ότι ε, δραστηριοποιούμεθα σε, σε διάφορου τομεί. Μετά, το θέμα της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, όπου τα κράτη-μέλη κάνουν αξιολογήσεις ομοτήμων. Πάλι η Κομισιόν ενθαρρύνει, προτείνει, προετοιμάζει όλο το, το υλικό, προετοιμάζει το δρόμο και στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής τα κράτη-μέλη κάνουν αξιολόγηση ομοτήμων. Αξιολογεί το ένα το, οικονομικό, το κοινωνικό σύστημα του άλλου. Και εκεί πραγματικά υπάρχει μια τεράστια δυναμική και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ξεμείνου και στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικής, ε, Κοινωνικής συγγνώμη, ε, Πολιτικής. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ουγγρική κυβέρνηση έχει εμπλακεί ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες. Μετά, συνεργαζόμαστε στενά με τον ΩΣΑ, του οποίου είναι μέλος η Ουγγαρία. Εγώ ήμουν στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στον ΟΣΑ με όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για την Ουγγαρία. Και η Κομισιόν, όπως και τα κράτη-μέλη, επικεντρώνεται κυρίως στον κοινωνικό αντίκτυπο της ε, κατάστασης μετά της χρηματοοικονομικής, ε, χρηματοπιστωτική, οικονομικής, πολιτικής κρίσης. Η Ουγγαρία είναι μια χώρα που δέχεται ιδιαίτερες ε, πιέσεις ε, οικονομικά. Το Μάιο του 2012 ξέρετε ότι η Ουγγαρία έχει μπει ε, σε πρόγραμμα ισοζυγίου πληρωμών όχι σε πλήρες πρόγραμμα αλλά έχει οθετήσει κάποια πολύ αυστηρά μέτρα που μάλλον αυτός είναι ένας από τους λόγους που η κυβέρνησή σας δεν ήθελε να εμπλακεί, να κάνει το phase in όπως λέμε σε, μια, έτσι, σε ένα βάθος χρόνου να υιοθετήσει αυτά τα μέτρα για τους πολίτες της. Οι, μεταρρυθμίσεις για τα συνταξιδοτικά συστήματα είναι πάντα δύσκολες, σε όποια χώρα και να γίνουν, σε όποια ήπειρο και να γίνουν. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ποτέ δεν είναι εύκολες. 18 κρατημέλη αυτή τη στιγμή κάνουν τέτοιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και η Κομισιόν παρακολουθεί και τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτών των διαδικασιών. Ανησυχούμε ιδιαιτέρως για την αυξανόμενη ένδια των εργαζόμενων σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς επίσης και για την ένδια των συνταξιούχων. Οπότε αυτή πραγματικά είναι, αυτός είναι ο πυρήνας των, ε, της ενασχόλησής μας. Ε, σας ακούμε, αλλά νομικά δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, πρέπει να σας θυμίσω ότι η διερμηνείς θα είναι μαζί μας μέχρι τις 6.30 και μας τελειώνει και ο χρόνος. Πρώτος που θέλει το λόγο, ο κύριος Ταμπάτσι. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν αρκετές χιλιάδες άτομα που ανησυχούν όταν βλέπουν αυτά που συμβαίνουν στην Ουγγαρία γιατί θίγονται τα δικαιώματά τους θέλουν να γνωρίζουν εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών θα τους βοηθήσουν. Γι' αυτό χρειάζεται μια υπεύθυνη απόφαση και κοινωνικά και ηθικά. Παρακαλώ, προσέξτε. Έχουμε τέσσερις βασικές αρχές που θίγονται. Ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υιοθετήθηκε το μέτρο αυτό στην Ουγγαρία. Πρώτα απ' όλα αυτός ο αναδρομικός χαρακτήρας του νόμου είναι αντίθετος με βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι θεμελιώδεις αρχές ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλά και διάφορα που θίγονται επαναλαμβάνω όπως και κεκτημένα δικαιώματα προηγούμενα κλπ. κλπ. Και τα έχει υπερασπιστεί αυτά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρακαλώ προσέξτε κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προσέφυγε στο δικαστήριο κατά της Ουγγαρίας όσον αφορά τη συνταξιοδότηση των ε, δικαστών από τα 70 χρόνια σεξιότητας πήγε στα 72 έτσι αυθαίρετα και είναι κάτι το παράνομο αυτό που συμβαίνει. Και αυτό ο αναδρομικός χαρακτήρας αυτού του μέτρου τώρα για τους Τουρκικούς είναι κάτι το απαράδεκτο. Και ακόμα από νομική πλευράς οι κοινωνικές παραχέ, εντάξει οποιαδήποτε στιγμή βλέπουμε ότι αφαιρούνται, καταπατούνται ε, και δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά δυνατότητα προσφυγής, διαμαρτυρίας προσφυγής. Δεν μπορούν να προσφύγουν σε δικαστήριο και να αμφισβητήσουν αυτό το μέτρο. Ούτε και στο Στρασβούργο πουθενά σε κανένα δικαστήριο. Και τώρα είναι η πρώτη φορά εδώ που μιλάνε για το πρόβλημά τους. Θέλουν να μπορούν να κάνουν μια προσφυγή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το εξετάσει αυτό γιατί στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν δικαιώματα, δηλαδή προσφυγή κατά μιας, καταδικαστική απόφαση. Επίση, καταδικαστικής απόφασης. Επίσης, ο σεβασμό τη ανθρώπινη αξιοπρέπειας. Αυτή η ε, εργάτες στα ορυχεία, από αστυνομικά σώματα, από στρατιωτικά σώματα, όλοι αυτοί, ε, όλα αυτά τα δικαιώματα καταπατούνται και είναι κατά της αξιοπρέπειάς τους. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά να ζητηθεί μια, η επίσημη άποψη της ε, Ουγγρικής κυβέρνησης και να έχουμε και τη σύσταση μιας ερευνητικής επιτροπής που να ζητήσει από εδώ, ναι, ξεκινώντας να σταματήσει πια να καταπατάει το νόμο και να αποζημιώσει μάλιστα και τα θύματα των μέτρων αυτών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στάση της και μάλιστα αμέσως. Ευχαριστώ. Thank you. Colleague Ο κύριος Μπουστινάρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριοι αναφέροντες, από την αρχή η απάντηση της ε, Κομισιόν δεν είναι απλώς ε, μη ικανοποιητική, αλλά είναι πολύ τεχνική, είναι κωδικοποιημένη. Όποτε συζητούμε θέματα πεπρωμένου, είναι πολύ γραφειοκρατική η απάντηση. Και το λέω αυτό γιατί η Κομισιόν μας λέει γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. και γιατί μπορούμε μόνο να δώσουμε απαντήσεις θεωρητικές σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Καταρχάς, τα κριτήρια της, Κοπενχάγη, της Κοπενχάγης ήταν προϋπόθεση για την πρόσβαση στην Ευρωπα... για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη. Στα κριτήρια της Κοπενχάγης και ε, στα διαπραγματευτικά πακέτα, όπως και για τη Ρουμανία, αλλά και για άλλες ε, χώρες, υπάρχει ένα κεφάλαιο για την, ε, το δικαστικό τομέα, το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητα του νομικού πλαισίου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Όλα έγιναν εν μία ανοιχτή, χωρίς να υπάρξει καμία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεύτερον, οι συντάξεις θεωρούνται στοιχείο ενεργητικού στη διάθεση της ε, κυβέρνησης. Αλλά είναι δικαίωμα ιδιοκτησίας. Και ως τέτοιο δεν μπορεί να παραβιάζεται. Τρίτον, η αρχή της αναδρομικής παρέμβασης δεν έχει λειτουργήσει από τον καιρό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατηρίας. Ε, λειτουργήσε μόνο σε απολυταρχικά θεστώτα. Πώς μπορεί η Κομισιόν λοιπόν να λέει ότι αυτή η αρχή της αναδρομικότητα θα γίνει ευρωπαϊκό α, κεκτημένο. Και επίση να ρωτήσω και τους αναφέροντες. Ίσως να έχω λανθασμένε εγώ πληροφορίε, αλλά ρωτώ. Έχετε λάβει κάποιο επίσημο έγγραφο με τους ε, νομικούς λόγους επί τη βάση των οποίων το δικαίωμα στη σύνταξη απερίφθη ή αφαιρέθηκε από αυτούς που το κατήχαν, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο επίσημο έγγραφο ή σημείωμα. Οπότε οι αναφέροντες απλώς σταμάτησαν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη πια. Ρωτώ λοιπόν, είναι δυνατόν να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα δικαστήρια για αυτούς τους αναφέροντες. Δεν είχαν κανένα ένδικο μέσο στα χέρια τους, στη χώρα τους ή αλλού. Γιατί δεν υπάρχει νομική εξήγηση, δεν υπάρχει νομικός λόγος που να λέει ότι από αύριο αυτό το δικαίωμα αφαιρείται από εσάς. Αν λοιπόν συνέβη αυτό, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα. Όταν παραβιάζονται, τι νόημα έχει να υπάρχουν αν είναι να τα παραβιάζουμε. Συνέχεια λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται από την κρίση. Στη Ρουμανία όμως η προηγούμενη κυβέρνηση προέβησε παρόμοια μέτρα και πήγε κάποιο, πήγαν αυτοί που τους έπληταν στα δικαστήρια και κέρδισαν τη δίκη γιατί όμως είχαν πρόσβαση στα δικαστήρια και η κυβέρνηση πρέπει τώρα να πληρώσει αυτή, η νυν κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει τα όσα έκανε η, παλιά, προηγούμενη κυβέρνηση. αυτό το βάρος μετακυλίεται στους, ε, στις μεταγενέστερες, στις μελλοντικές κυβερνήσεις. Και τώρα η Κομισιόν μας λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ε, αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν εμέσως δέχεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται από το κοινωνικό μοντέλο που έχει υποστηριχθεί από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν λένε στους στρατιωτικούς που υπηρέτησαν την πατρίδα τους και θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα τους ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτούς. Κατά συνέπεια προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά δεύτερον. Η πρόεδρος της Επιτροπής μας να ε, κοινοποιήσει, να ενημερώσει την ε, Ουγγρική κυβέρνηση και να ζητήσει εξήγηση και να ζητήσει το, νομικό, την νομική επιχειρηματολογία βάσει της οποίας απαγορεύεται η πρόσβαση στην δικαιοσύνη για αυτούς τους αναφέροντες. Η Επιτροπή Επασχόλησης επίσης θα πρέπει να παρέμβει σε αυτό το θέμα. Και τέλος, να στείλουμε ένα μνημόνιο στον Επίτροπο Άντορ, που παρόλο που είναι Ούγγρος, δεσμεύεται από τα καθήκοντά του να πει, να απαντήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν μπορούμε να καταδικάσουμε 40.000 Ούγγρους πολίτες στην φτώχεια μετά τόσα χρόνια ε, υπηρεσίας προς την πατρίδα τους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι ο χρόνος περνάει. Οπότε παρακαλώ αν έχετε κάτι καινούριο να προσθέσετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν ικανοποιητική η γνωμοδότηση. Μιλάμε για 40.000 πολίτες. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί για, για αυτούς. Όταν μιλήσαμε για, για άτομα που έχουν ε, μπει στη σύνταξη λόγω προβλημάτων αναπηρίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε, είπε ότι, ότι είναι απαράδεκτο το να μην υπάρχει μεταβατική περίοδος. Αυτό είναι μη αποδεκτό το Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είπε ότι υπάρχει μια προτεραιότητα εδώ υπάρχει μια πιθανότητα από την Επιτροπή να αγγίξει αυτό το θέμα. Ελέγχθη ελέγχθη ότι τα άτομα για τα οποία μιλήσαμε το πρωί και, και αυτοί 40.000 υπάρχει δυνατότητα προσφυγές ε, ε το αρνήθηκαν κάποιοι αυτό αλλά η βάση στο ευρωπαϊκό δίκαιο λέει ότι έχει κάνει αυτό δικαίωμα προσφυγής. Θα πρέπει να ζητηθεί κάτι πάνω σε αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να το δούμε. Ευχαριστώ. Να σας δώσω το λόγο εσάς πρώτα, κύριε Πάκο. Όχι, όχι, όχι, όχι εσείς πρώτα, περιμένετε. Μισό λεπτό, πρώτα, πρώτα εσάς και πρώτα εσείς και μετά εσείς, συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώς, θα, πώς εξελίσσεται σήμερα ο διάλογος και ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό διάλογο που κρύβει ένα τεχνικό. Όλοι το ξέρουν. Έχουμε μια ε, ένωση 3.000 ατόπων με 1860 υπογραφές. Η ελέγχθη ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες άτομα τα οποία παρακολουθούν στο διαδίκτυο αυτό, αυτή τη συζήτηση. Όλοι στην Ουγγαρία ξέρουν ότι αυτό είναι πολιτικό θέμα. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι το σύστημα το οποίο υπήρχε στη Ουγγαρία και όπως δούλεψε δεν ήταν ένα σωστό σύστημα. Εμείς δεν είμαστε τώρα μια επιτροπή έρευνας για την Ουγγρική κυβέρνηση και επειδή αναφέρθηκε το θέμα της προσφυγής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εδώ είμαστε στη, σε μια επιτροπή που ασχολείται με τις αναφορές και πρέπει να αποφανθούμε αν είμαστε οι αρμόδιοι πάνω σε αυτό το θέμα ή όχι. Το ότι δεν γνωρίζουμε το δίκαιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να, σεβαστούμε, να το σεβαστούμε. Είναι εδώ αυτό ένα θέμα πάνω στο οποίο η Επιτροπή μας δεν έχει αρμοδιότητες. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν θα επαναλάβω. και τα οποία μας κάνουν ένα μήνυμα σε σίγουροι αν έχουν καταστρατηθεί ε, το, αν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μπορεί, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πολλά άλλα δικαστηρία, αλλά δεν είναι η Επιτροπή Αναφερών αυτή, αυτή η οποία θα αποφασίσει. Θα είμαι σύντομος και θα επανέλθω αν χρειαστεί. Εγώ στην Αυστρία ήμουνα γενικός ε, γραμματέας μιας μεγάλης ένωσης ε, συνταξιούχων που είχε πλήρες, ε, πλήρη δυνατότητα παρέμβαση ως, ε, ως ε, κοινωνικός εταίρος. Δηλαδή κάθε φορά, κάθε χρόνο διαπραγματευόμασταν από κοινού με την κυβέρνηση της συντάξης. Ξέρουμε επακριβώς από τη δική μας την κυβέρνηση και από όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις ότι τα ευρωπαϊκά κρατημέλη έχουν εμποδίσει με κάθε τρόπο να υπάρξει νομοθετική αρμοδιότητα για θέματα ε, συντάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν την κατανόηση σας όταν λέω ότι εμείς ας είμαστε ε, ειλικρινεί απέναντι στους αναφέροντες με το πρόβλημα που έχουν. Ας μην τους δημιουργούμε ελπίδες ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί κάτι να γίνει. Εγώ ζητώ λοιπόν να υπάρξει σωστή στοχοθέτηση, να δούμε ποιες είναι οι διάφορες επιλογές εκτός τούτης της ομάδας, είτε είναι ε, το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε είναι πολιτικές επαφές μέσω των επιτρόπων, όλα θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε αυτό το στόχο έτσι ώστε αυτό το επίπεδο το ευρωπαϊκό να καταφέρει κάτι γιατί θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμβάλει ε, ε, ουσιαστικά. Αύριο θα ψηφίσουμε τη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις, το πρώτο μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένωσης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό όχι για να είμαι αρνητικός, αλλά για να μην δημιουργούμε ψευδείς ελπίδες και φρούδες ελπίδες στους ανθρώπους αυτούς. Παρακαλώ λοιπόν την ε, κατανόησή σας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά να σας πω ότι εδώ μιλούμε για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Αναφορών πάντα ε, ενεργώς ε, παρενέβαινε σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κλείνοντας λοιπόν, για να κάνουμε έτσι μια περίληψη των διαφόρων θέσεων, θα, θα διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Δεύτερον, θα ζητήσουμε περισσότερες εξηγήσεις από την Κομισιόν για το γιατί δεν μπορεί να γίνει το α, β και το γ και θέλουμε κάτι γραπτός. Και τρίτον, να ζητήσουμε μια επίσημη θέση από την Ουγγρική κυβέρνηση και να δούμε τι θα μας απαντήσουν, πώς θα μας εξηγήσουν αυτοί οι ίδιοι την κατάσταση. Και μετά η ε, Γραμματεία θα συλλέξει τις απαντήσεις και θα συνεχίσουμε στην Επιτροπή τη συζήτηση, εάν αυτό σας βρίσκει σύμφωνος, συνάδελφοι. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν τους αναφέροντες για την ε, παρουσίασή τους, για την προσπάθεια που έκαναν. Και συνεχίζουμε με το σημείο 19. Αναφορά 1557 του 2009. Νομίζω ότι είναι παρόντες οι αναφέροντες. Α, όχι, μόνο η Κομισιόν είναι η παρούσα. Εντάξει. Παρακαλώ η Κομισιόν να πάρει το λόγο. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ οι ε, αναφέροντες, οπότε θα ήθελα να κάνω μια περίληψη ε, των όσων υπόθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής Αναφορών. Λάβαμε ένα έγγραφο από την Ουγγρική Κυβέρνηση που εξηγεί τις απόψεις τους για την αναφορά και τις τελευταίες μέρες λάβαμε και την ε, απάντηση από την αναφέρουσα. Ελέγχοντας τις απαντήσεις της Ουγγρικής κυβέρνησης, εξεκολουθούμε να μένουμε στη θέση μας ότι δεν υπάρχει απόδειξη που να δείχνει ότι υπάρχει παραβίαση του της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Υπήρχε ένας μακροσκελής κατάλογος στην ε, απάντηση με πολλές εξηγήσει για τα νέα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρετε ότι η αναφορά υπευλήθη όσο ήταν στην εξουσία η προηγούμενη κυβέρνηση. Η αναφέρουσα στην απάντησή τη, λέει ότι ένα από του λόγου ε, για το ότι υπευλήθησαν οι αναφορά του 2009 είναι ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να διαπραγματευτεί με εκπροσώπου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λέει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί μετά την αλλαγή τη κυβέρνηση και τώρα καλούνται σε συνεδριάσεις και λαμβάνονται υπόψη οι απόψει τους. Οπότε κάποια από τα προβλήματα που αναφέρονται στην αναφορά έχουν λυθεί. Εμείς λέμε ότι η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να, ε, κάνει, να ξεκινήσει τη διαδικασία παραβάση. Είναι το ίδιο με την προηγούμενη αναφορά ως προς αυτό. Υπάρχουν θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και αναφέρουσα λέει ότι το βασικό πρόβλημα ε, για το είναι το εμπορικό περιβάλλον στην Ουγγαρία. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά το τι κάνει η κυβέρνηση και στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα είμαστε σε επαφή με την Ουγγρική Κυβέρνηση. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, όπως λέει και η αναφορά, ήδη έχει ε, υποβάλει ένα έγγραφο πολιτικής για το σχέδιο δράσης που καταγράφει διάφορες συστάσεις προς την αγγλική κυβέρνηση ώστε να δημιουργήσει ένα επωφελές για τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Να δώσω το λόγο και σε έναν από τους συναδέλφους για τα θέματα φορολογίας που αναφέρονται στην αναφορά. Πολύ σύντομα όμως. Η αίσθηση της Γενικής Διεύθυνσης Ταξούτ που εκπροσωπώ είναι ότι ε, η αναφέρουσα γνωρίζει ότι την ε, κριτική που έχει ε, αναφέρει, που έχει παρουσιάσει απέναντι στην εθνική φορολογική πολιτική. Υπάρχει βεβαίως και η οδηγία για τον ΦΠΑ που προτείνει ένα εναρμονισμένο σύστημα ΦΠΑ και βεβαίω ε, δεν υπάρχει παραβίαση, το επιβεβαιώνω. Η υποχρέωση καταβολή του ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το αν έχει πληρωθεί το τιμολόγιο, ε, ε, προβλέπεται από την σχετική οδηγία. Πρέπει να πω όμω ότι υπάρχει επιλογή για τα κράτη-μέλη να επιλέξουν και άλλο σύστημα. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 66. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ο ΦΠΑ αφαιρείται όταν έχει ληφθεί η πληρωμή. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση για το πρόβλημα της αναφέρουσας, αλλά αυτό δεν είναι υποχρέωση για τα κράτη-μέλη, είναι επιλογή τους, που θα πρέπει να τη μελετήσουν τα ίδια, η ε, Ουγγαρία προκειμένου. Επίση, μια υπηρεσία όταν παρέχεται ή όταν γίνονται κάποια έργα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, δεν έχουν εξοφληθεί, υπάρχει δυνατότητα να προσαρμοστεί η ε, φορολογική βάση. Αυτό μπορούν τα οποια δεν εχουν πληρωθει δεν εχουν εξοφληθει υπαρχει δυνατοτητα να προσαρμοστει η φορολογικη βαση αυτο μπορουν τα μελη να το κάνουν στα πλαίσια του άρθρου 92, παράγραφος 2. Παρόλα αυτά, η Ουγγαρία για τους δικούς της πολιτικούς λόγους ή για λόγους φορολογικής πολιτικής δεν έχει επιλέξει αυτή την άγουσα. Τώρα για το χρονικό όριο για την ε, ε, επιστροφή του ΦΠΑ, το άρθρο 186 της οδηγίας για το ΦΠΑ προβλέπει ε, προτείνει στα κράτη-μέλη να ορίσουν τι ε, συνθήκε κατά από τι οποίε θα γίνει αυτή η ε, επιστροφή. Δεν είναι λοιπόν ορμονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα αυτό. Και μετά από διαρεύνηση του ουγγρικού συστήματος είδαμε ότι υπάρχει αποζημίωση, επιστροφή μετά από 75 μέρες και μετά από 30 ή 40 μέρες όταν δεν έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο. Αυτό νομίζω ότι συνάδει με περισσότερες πρακτικές και από άλλα κράτη-μέλη, επομένως δεν υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σημερίζουμε λοιπόν τα, τις των ε, μικρομεσών επιχειρήσεων, αλλά η πίεση πρέπει να ασκηθεί στην ε, Ουγγρική κυβέρνηση, γιατί η νομοθεσία του ε, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επομένω δεν μπορεί να κάνει κάτι η Κομισιόν. Ωραία, σα ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει μείνει κανένα συνάδελφο στην αίθουσα, οπότε θα παρακολουθούμε την ε, αναφορά και θα την κλείσουμε κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Σα ευχαριστώ όλου που ήσασταν παρόντε. Η πρόεδρο ευχαριστεί και του και εμείς. Πέρα συνεδρίασης. Καλό σας βράδυ.